Could people please take their seats? Μπορείτε να καθίσετε παρακαλώ. Πότε δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω αυτό το σφυρί, αλλά τώρα θα αρχίσω. I've got two teenage sons. <laughs> <laughs> Oh dear, thank you very much. Please can you take a seat? There's still some of the advisors at the back of the room. Thank you very much. Κάποια πηγαδάκια αν μπορούν να διαλυθούν στο πίσω μέρος της αίθουσας. Ήταν εργόδες το πρωί κύριε Επίτροπε. Αλλά με μεγάλη χαρά ξαναγυρνάμε στην Επιτροπή εσωτερικής αγοράς και με μεγάλη χαρά χαιρετίζουμε και καλωσορίζουμε τον κύριο Άνσιπ, ένα παλιό φίλο, να μας ενημερώσει για τα θέματα που ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας. Ε, κανονικά την ε, πέμπτη το απόγευμα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη προσέλευση. Έχουν έρθει όλοι αυτοί για να σας ακούσουν. Ξέρω Κάποιοι πρέπει να φύγουν να προλάβουν τα αεροπλάνα τους. Και γι' αυτό είμαστε απόλυτα έτοιμοι να ακούσουμε τι θα μας πείτε. Από τότε που είχαμε ξανασυναντηθεί έχουμε δει ορισμένα ψήγματα από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων που περιμένουμε από εσά, αλλά περιμένουμε να μας πείτε αυτά που είναι οι προθέσεις σας για την εσωτερική αγορά θα λάβει λοιπόν το λόγο ο κύριος Επίτροπος και μετά θα έχουμε χρόνο για ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων. Βλέπω και άλλους να έρχονται. Καθίστε παρακαλώ εσείς που συνοθήσετε στην είσοδο. speech or just points Λοιπόν, θα θέλαμε να σας ακούσουμε, λέει η Πρόεδρος, και μετά θα ακολουθήσουν τα ερωτήματα. Παρακαλώ. Κάθε φορά που μιλάτε μας λέτε και καινούργια πράγματα. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρος, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά είμαι πάλι μαζί σας στην αρχή της εντολής μου είπα θα προσπαθήσω να κρατήσω στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσω να σας παρουσιάσω ποιες είναι οι προτεραιότητες της ε, ψηφιακής ενίας αγοράς ε, και σε... σε σχέση με αυτό είναι φανερό ότι η Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι θέλουν περισσότερη επιλογή, πιο ανταγωνιστικές τιμές και τη δυνατότητα να απολαμβάνουν όλο αυτό των προϊόντων. Η ψηφιακή αγορά αφορά επίση επιχειρήσεις, είτε είναι καινοτόμε, ε, startups ή παραδοσιακές βιομηχανίες. Στην ψηφιακή αυτή εποχή θα πρέπει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβουμε υπόψη αυτήν την τεράστια αγορά 500 εκατομμυρίων πελατών. Η παραδοσιακες βιομηχανιε στην ψηφιακη αυτη εποχη θα πρεπει μεσα στην ευρωπαικη ενωση να λαβουμε υποψη αυτην την τεραστια αγορα 500 εκατομμυριων πελατων η στρατηγικη μας θα βασιστεί σε τρεις πυλώνες πολιτικής που έχουν σε στόχο να απελευθερώσουν το δυναμικό της ψηφιακής οικονομίας και το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης. Για να γίνει αυτό το όραμα πραγματικότητα και να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το επιγραμμικό περιβάλλον, θα πρέπει να τονίσουμε ορισμένες ε, προτεραιότητες. Να μην υπάρχει άρνηση πρόσβαση σε ιστοσελίδες επί τη βάση γεωγραφικής προέλευσης και αποκλεισμού, παραδείγματος χάρη. Μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα με το να άρουμε τους φραγμούς. Σκεφτείτε το υψηλό κόστος της διαμεθοριακής παράδοσης δεμάτων, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για αυτούς που ψωνίζουν στο διαδίκτυο και εμποδίζει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη. Ή, αν δείτε την, τον γεωαποκλεισμό στο geo-blocking, που ακριβώς αυτό ανέφερα προηγουμένως, τον αποκλεισμό από ιστοσελίδες λόγω του τόπου που βρίσκεται κανείς. Δεν έχει νόημα να υπάρχει τέτοιο εμπόδιο για πρόσβαση σε ιστοσελίδες. Είναι μια πρακτική που όχι μόνο είναι εμπόδιο για το εμπόδιο, αλλά αντίκειται στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ενίας Αγοράς. Οι καταναλωτές θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο αν, μπορούν, αν θα μπορούσαν να επιλέξουν αγαθά και υπηρεσίες από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ψωνίζουν στο διαδίκτυο. Πολλοί από τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν καταναλωτές και οι επιχειρήσεις σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας κατακαιρματισμένης αγοράς. Έχουμε διαφορετικούς εθνικούς κανόνες στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <clears throat> κανόνες για αγορές στο διαδίκτυο και ψηφιακές υπηρεσίες, όλα αυτά είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα όπως και οι κανόνες για την προστασία των καταναλωτών και για τον νόμο για συμβάσεις. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, υπάρχουν πολλές ε, διαφορετικές πρακτικές για τις εταιρείε στο διαδίκτυο χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά δημιουργούν μία οπιστέλκουσα στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Αυτό αποθαρρύνει τους επενδυτές και χρειαζόμαστε περισσότερους επενδυτές στον ψηφιακό κόσμο. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή και λειτουργική υποδομή για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα αυτά, όπως και ένα σωστό κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει να ε, άρουμε όλους αυτούς τους φραγμούς που δεν μας επιτρέπουν να εκμεταλλευτούμε πλήρως μια ευρωπαϊκή αγορά για τηλεπικοινωνίες να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα για τις ε, τηλεπικοινωνίες και τις ε, εταιρείε του διαδικτύου. Να προωθήσουμε την επένδυση και την καινοτομία και να εξασφαλίσουμε ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε υψηλή ταχύτητα σε ευρυζωνικά δίκτυα. Κυρίε και κύριοι, για μένα είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, προς μια πραγματική ενιαία αγορά για τον επιγραμμικό <clears throat> χώρο, χωρίς προηγουμένως να κάνουμε κάποια αλλαγή στους κανόνες της αγοράς και να επιτύχουμε τη ε, σωστή, εφαρμογή ψηφιακής υποδομής. Αλλά και οι στρατηγικές μας θα πρέπει να υπερβούν αυτό το σημείο. Θα πρέπει να προσβλέψουμε προς ένα μέλλον ψηφιακό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προετοιμάσουμε για νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, καθώς ο κόσμος μας προχωρεί σε χώρους όπως είναι το υπολογιστικό δίκτυο, το διαδίκτυο των αντικειμένων και η ταχεία ανάπτυξη των δεδομένων. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να θέσουμε τις βάσεις για μια στεναρή ανάπτυξη στο μέλλον, ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να λάβει πλήρως υπόψη της και να εκμεταλλευτεί την ψηφιακή οικονομία, όπου τα δεδομένα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία και όπου οι άνθρωποι έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα και να είναι στον κυβερνόχωρο με απόλυτη εμπιστοσύνη. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό για όλα αυτά. Φανταστείτε τα θέματα αυτοματοποίησης, της βιώσιμης και καθαρής διαδικασίας παραγωγής κτλ. Το να ενσωματώσουμε πλήρως την πληροφορική στη διαδικασία παραγωγής, αυτό θα είναι απαραίτητο για να μπορέσει η Ευρώπη να διατηρήσει την ισχυρή βιομηχανική της βάση. Μέχρι τώρα η ψηφιοποίηση της ε, βιομηχανίας και των επιχειρήσεων στην Ευρώπη έχει καθυστερήσει. Πρέπει να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Χρειαζόμαστε κοινά πρότυπα και διαλειτουργικότητα. Όλα αυτά είναι κέρια για την Ευρώπη και στο πλαίσιο της πρόθεσης περισσότερων υπηρεσιών στην ε, ευρωπαϊκή κοινωνία και ε, περισσότερης παροχής δημοσίων υπηρεσιών και διοίκησης σε επιγραμμικό επίπεδο. Οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν παραγωγικά να γίνουν πιο γρήγορες, πιο αποτελεσματικές, πιο βολικές και επίσης να εξοικονομήσουν τα χρήματα των πολιτών. Γι' αυτό οι δημόσιες υπηρεσίες διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη στρατηγική της ψηφιακής ενίας αγοράς. Μπορούμε λοιπόν να θέσουμε σε εφαρμογή αυτήν την αρχή του να έχουμε ενιαία πρότυπα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε 5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Γιατί λοιπόν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες θα πρέπει να υποβάλουν τις ίδιες πληροφορίες πάλι και πάλι εκ νέου και ξανά στις ίδιες υπηρεσίες ή τουλάχιστον στην ίδια υπηρεσία πολλές φορές όταν αυτά τα στοιχεία μπορούν να υπάρχουν μία φορά και για πάντα. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν με την ενιαία ψηφιακή αγορά μπορούμε να καλύψουμε πολλούς χώρους του επιχειρήν Μπορούμε έτσι να βελτιώσουμε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Η ψηφιακή αγορά και η στρατηγική της ψηφιακής αγοράς θα πρέπει να ατενιστεί και μια, ως μια ευκαιρία για τα επόμενα χρόνια και η κοινή μας συνεργασία ξεκινάει όπως ανέφερα προηγουμένως στις 6 Μαΐου. Είμαι έτοιμος να απαντήσω στα ερωτήματά σας λοιπόν. Ευχαριστώ. Oh, um, uh, Η πρόεδρος. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε τις αγορεύσεις, καλώς ήρθαν οι προσκεκλημένοι. Είναι κάποιοι φοιτητέ, σπουδαστέ από Ιταλία, Πολωνία, Σλοβακία και Κροατία βάσει του προγράμματος ε, ανταλλαγών. Χρειαζόμαστε περισσότερου νέου να εμπλέκονται στην πολιτική. Ήρθαν ακριβώ στην κατάλληλη στιγμή. Περισσότερου αναγκαίε, περισσότερου νέου. Ε, τώρα είχαμε τον ε, αντιπρόεδρο Άνσεπ, ξέρετε, που μα μιλά για τα θέματα της ψηφιακής ενία αγοράς για να δούμε γιατί χρειαζόμαστε περισσότερες τέτοιες προτάσεις για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει την πρόκληση η Ευρώπη για την ε, ψηφιακή εποχή. Από ό,τι βλέπω πάρα πολύ από εσά ήδη επικοινωνείτε ε, με την πατρίδα σας ψηφιακά. Και, να, τέτοια ανταλλαγή απόψεων ελπίζουμε ότι θα δώσει απαντήσεις και κάποιες ερωτήσεις πριν καταλήξουμε σε επίσημες προτάσεις. Οπότε τώρα για να δούμε, ε, βάσει των όσων έχουν καταγραφεί ως ε, αγοραστές, τρεις-τρεις, ε, λοιπόν η πρώτη τριάδα συναδελφών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και στον Επίτροπο. Να περιμένω μέχρι να βάλετε τα ακουστικά σας. Um, okay. just Η Πρόεδρος, αν θέλετε να βάλετε τα ακουστικά σας στα διαφορετικά κανάλια, θα ακούτε τις διάφορες γλώσσες. Μπορείτε να βρείτε και τη δική σας γλώσσα. Να βρείτε το κανάλι σας. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ, Επίτροπε, για την παρουσίαση των όσων μπορούμε να περιμένουμε για το μέλλον. Νομίζω ότι θίξατε κάποια πολύ σημαντικά θέματα στα εισαγωγικά σας σχόλια, τα οποία μας ε, απασχολούν ιδιαίτερα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αφενός πρόκειται για τα πολλά εμπόδια, τα πολλά προσκόμματα της εσωτερικής αγοράς, τα οποία και δεν επιτρέπουν να μοιραστούμε τα επιτεύγματα της ψηφιακή αγοράς. Να ωφεληθούν όλοι οι καταναλωτές. Και η δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν λειτουργεί καλά το ζήτημα, η ενιαία αγορά, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης από πλευρά των πολιτών, γιατί είναι πολύ διαφορετικοί οι κανόνες στα κράτη-μέλη και δεν έχουμε ουσιαστικά πραγματική επισκόπηση. Θα ήθελα λοιπόν να κοιτάξουμε αυτή η ενιαία αγορά πώς πρέπει να ρυθμιστεί στο μέλλον, με βάση ποιες αρχές, ξέρετε. Ότι υπάρχει μία παράδοση εναρμόνισης στην Ευρώπη και με την ε, οδηγία για την προστασία των καταναλωτών προσπαθήσαμε να πετύχουμε την πλήρη εναρμόνιση. Πιστεύω ότι είναι ο σωστός τρόπος αυτός ε, να προχωρήσουμε, γιατί και για τις επιχειρήσεις ε, και για τον πολίτη είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος. Θέλετε λοιπόν να αλλάξει αυτό. Θυμάμαι την ομιλία σας στις 26 Νοεμβρίου στην Ολομέλεια. Όταν είπατε ότι η αρχή της χώρας προέλευσης ε, πρέπει να αποτελεί τη βάση για την προστασία του καταναλωτή και για τις online, τις επιγραμμικές υπηρεσίες. Και τότε είχαμε πει ότι ε, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που θα προέκυπταν και ότι η ομάδα μου δεν συμφωνούσε. Για παράδειγμα, η αρχή της χώρας προέλευσης σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν 28 χώρες μέλη με διαφορετικές νομοθεσίες, τις οποίες θα εκμεταλλεύονται οι επιχειρήσεις. Και αυτό τι σημαίνει, την προστασία του καταναλωτή. Δεν θα είναι η υψηλότερη δυνατή. Ποια οδό λοιπόν θέλετε να ακολουθήσετε. Ελπίζω να το έχετε σκεφτεί καλύτερα. Και να προτίθεστε να συνεχίσετε στην οδό της πλήρους αρμόνισης. γιατί μόνο με κινήσει νομοθεσία και ρύθμιση θα μπορέσουμε στην Ευρώπη πραγματικά να καταργήσουμε όλα τα εμπόδια που υπάρχουν και πραγματικά ανυπομονώ να ακούσω την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κάλλας, ευχαριστώ πάρα πολύ και πολύ μπαίνω στον πειρασμό να σας μιλήσω στα εσθονικά. Um, I will just uh, do it in English, Όχι, όχι, θα μιλήσω αγγλικά για να είναι πιο εύκολη παρακολούθηση. Σήμερα οι γραμμές μετά, τα διαφορετικά μεταξύ του online και offline κόσμου είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν και είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε τις υπηρεσίες online από τις υπηρεσίες offline. Ελπίζω λοιπόν ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά να μην αγγίζει μόνο την ψηφιακή διάσταση αλλά και τους άλλους τομείς της οικονομίας Πολλά ερωτήματα έχω, μόνο κάποια εξ αυτών θα θέσω. Μιλήσατε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, διαχείριση. Και είπατε πόσο υστερεί εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, πρόκειται να συμβεί κάτι. Γρήγορα μάλιστα, προκειμένου να έχουμε κάτι να επιδείξουμε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην ε, Ευρώπη. Άλλο ερώτημα για, την, για τις πλατφόρμες, τις επιγραμμικές πλατφόρμες. Κοιτώντας αυτές τις πλατφόρμες online, εδώ δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης, ανάπτυξη. Αν και από ό,τι βλέπουμε στις συζητήσεις, το θέμα είναι μόνο πώς θα ρυθμιστούν αυτές οι πλατφόρμες, προκειμένου να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού με τις, με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Πώς λοιπόν θα διασφαλίσουμε ότι οι κανονισμοί και η ρύθμιση δεν παρεμποδίζουν την καινοτομία, το δυναμικό καινοτομίας. Μία άλλη ερώτηση για την βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για τις ε, εταιρείες ιδιαίτερα για τις ε, συστατήσει, τις νεοφυεί. Θα μείνει αυτό στην ε, στρατηγική ενιαία αγοράς ή θα υπάρχει και στην ενιαία αγορά τέτοια ρύθμιση για τι νεοφυεί. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε που ήρθατε σήμερα εδώ. Εντάχει σε συνέχεια τον είπε η Ευλήν να σας πω κάτι για την προστασία των καταναλωτών. Πολλές προσδοκίες αλλά και πολλά ερωτηματικά. Αυτό για το δίκαιο των πωλήσεων εγκαταλείφθηκε ως ιδέα αλλά θα πρέπει να δούμε τελικά τι απέμεινε από αυτή την πρόταση. Μήπως πρέπει να έχουμε πιο προχωρημένη εναρμόνιση ε, πέραν του κανόνα του δικαίου του, της χώρας του πολιτείου. Οπότε μήπως θα πρέπει να είναι σημείο αναφορά στη σύμβαση πολίσεως ο καταναλωτής και όχι ο πολιτής. Επίσης, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ιδίως όσον αφορά τις επιχείρησεις. γίνει Διάφορε ρυθμίσει για την ενιαία θηρίδα στα πλαίσια τη οδηγίας και της υπηρεσίας, για την ε, αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών ε, δεξιοτήτων και προσόντων. Οπότε μπορεί κανεί έτσι ηλεκτρονικά να μπορεί να έχει πρόσβαση για την προσ... Ε, για αυτέ τις πληροφορίες αλλά όλα αυτά τώρα είναι άνισας μεταξύ των κρατών μελών. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς θα υπάρξει μια υλοποίηση και εφαρμογή πλήρης, αποτελεσματική και κατά δίκιο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών για αυτές τις δύο οδηγίες. Μήπως θέλετε να επεκτείνετε την χρήση αυτών των δύο εργαλείων που σίγουρα θα τονώσουν τις οικονομικές αλλαγές στις δύο συνοριακές στην Ένωση. Α, τώρα μας έχουμε άλλους που έχουν εγγραφεί που είναι πολύ περισσότεροι. Οπότε πρώτα πρώτα μήπως ο κ. Συνεπρόεδρος μπορεί να απαντήσει. Dan Dalton, Ivan Stefanich, Emma McClarkin, Catherine Styler, Ava Paunova, Ava Paunova. Okay. Aldemosa. Anybody else? Κάποιος άλλος? Α, εντάξει. Ζητώ συγγνώμη γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσω να, έχω μάτια παντού σε αυτήν την αίθουσα. Κύριε Αντιπρόεδρε, θέλετε να απαντήσετε σε αυτούς τους τρεις και μετά να προχωρήσουμε. από εσάς ξατάτε, λέει ο Αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Πρώτα απ' όλα τα δικαιώματα των καταναλωτών. Όταν μιλούσαμε για την αρχή της χώρας προέλευσης, και το τι άλλαξε με την περίφημη πια εκείνη οδηγία είναι το ότι θέλαμε να προχωρήσουμε στην ε, πρόταση του καταναλωτή με τις ρυθμίσεις και με τον ΦΠΑ οπότε και έγινε αυτή η αλλαγή όσον αφορά την αρχή της χώρας προέλευσης και τώρα έχουμε την αρχή της χώρας του προορισμού όμως οι επιχειρηματίες λένε ότι είναι φραγμός η κατάτμιση της ευρωπαϊκής αγοράς. Αλλά και οι καταναλωτές παραπονιούνται για την πολυνομία των οργανισμών που προστατεύουν τα συμφέροντά τους. Σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να κάνουν μια αγορά γιατί οι πολιτές δεν διευκολύνονται να πληρώσουν, να πωλήσουν συγγνώμη προς την χώρα του καταναλωτή. Δεν ξέρουν το ρυθμιστικό πλαίσιο, δεν ξέρουν τι ισχύει εκεί. Και τώρα για το ψηφιακό περιεχόμενο. Εμεί θέλουμε να υπάρξει πλήρη αρμόνιση των κανονισμών, γιατί πρόκειται ακόμα για παρθένο έδαφος. Δεν έχουμε κανένα κανονισμό σε επίπεδο ένωσης γι' αυτά. Μα ούτε και σε εθνικό επίπεδο δεν έχουμε κάποια ρύθμιση. Τόσο αφορά για τα υλικά αγαθά και εμπορεύματα. Μπορεί να γίνουν αγορές και πωλήσει μέσω ίντερνετ. Και μπορεί να φτιάξουμε κάποιο είδου ενοχικό δίκαιο για αυτές. Είπαμε, δεν έπιασε τόπο το να κάνουμε ένα δίκαιο πολύ πανευρωπαϊκό. Προσέχουσε και στο κοινοβούλιο. Αλλά να έχουμε κάποια ενημέρωση με τον κανονισμό και ελπίζουμε ότι θα καταστεί έτσι ευκολότερο να συνελάσσονται οι εταιρείε διασυνοριακά. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να ρωτήσατε επίσης. Η απάντηση είναι ναι. Έχουμε τώρα μια σωρία παραδειγμάτων και περιπτώσεων. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλα τα κρατη ουσιαστικά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι υπηρεσίες και αυτά τα παραδείγματα δεν ωφελούν. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διασυνοριακά. Δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα. Πρέπει να βρούμε λύση αυτά τα προβλήματα και στα πλαίσια της στατικής για μια ενιαία ψηφιακή αγορά. Έχουμε την οδηγία που αποκαλείται η Άιντας και αμοιβή αναγνώριση των ψηφιακών ταυτοτήτων. Και όταν αυτή η οδηγία ή άιντας πλήρως εφαρμοστεί, ε, τότε θα υπάρχει πρόσβαση διασυνοριακά. Ναι. Και όσον αφορά τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την τεχνική διακυβέρνηση. Όμως, ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και τα πράγματα δεν θα είναι τόσο ρόδινα, εύκολα. οι Ιντερνετικές πλατφόρμες έχουν μέλλον. Και μιλώ και για την συμμετοχή σε αυτές. Γιατί αρέσουν στον κόσμο. Είναι θέμα αποτελεσματικότητας που έχουμε. Και ενώ τώρα για κάποιες πλατφόρμες φορολογικών υπηρεσιών, δεν θέλω να ονομάσω αυτές τις εταιρείες είναι μόνο ένας επίτροπος δικαιούται να σας τα πει συγκεκριμένα, δηλαδή μία επιτροπή, κύριε Βέσταγκερ, για πολιτικές. Όπως είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Έτσι είναι η κατάσταση σήμερα στον τραπεζικό τομέα. Όχι γιατί οι τράπεζες Καλά καλά δεν σα είπα για ποια εταιρεία απλώ Ξεχάστε το απλώς. Απλώς σας παρέθεσα τι είπε εκείνο. Έχουν ζημία στου πιο επικερδείς τομεί των Ιντερνετικών πλατφόρμων. οι οποίες όλες τους και όλοι οι υπάρχοι υπηρεσιών πρέπει να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς μας. Δεν μπορεί κανείς να τους παρακάμψει. Όμως, αυτές οι πλατφόρμες πρέπει να υποστηριχθούν, γιατί είναι πραγματικά αποτελεσματικές. Και είναι καλές υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν στον κόσμο. Οι οποίοι όμως άνθρωποι που απολάβουν των υπηρεσιών παραπονούνται. Ας πούμε για τις μηχανές αναζήτησης. Όπως σας είπα, Πολλέ φορές δεν πειράζει. Κάποιες εταιρείε έχουν δεσπόζουσα θέση. Ακόμα και μονοπωλιακή. Αλλά κανείς δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί και να καταχραστεί αυτής της δεσποζούς θέσεως. Όταν δεν υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις και αμφιβολίες για κάποιες πλατφόρμες, ότι δηλαδή αυτό καταχρώνται τη δεσποζούς θέσεως ότι παραβιάζουν κάποιο κανονισμό, τότε ερευνούμε και παρεμβαίνουμε. Φυσικό είναι. Σε συνέχεια για τις μηχανές αναζήτησης. Τι είναι με τις επαμοιβή που προσφέρουν για το αποτέλεσμα και τις κάθε έρευνες. Παρέχουν και άλλες υπηρεσίες. Και, και τελικά ποιοι είναι πρωτοπόροι στην αγορά. Επομένως είχαμε εκείνη την πρόταση σχετικά που απεκρούσε από το Κοινοβούλιο. Άρα δεν συνεχίσουμε αυτήν την κατεύθυνση. Αυτά. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρο. Πρώτα περάσουμε στο επόμενο θέμα, στην ε, προστασία των καταναλωτών, γιατί είμαστε και αρμόδιοι για θέματα προστασία των καταναλωτών. Και διαπιστώνω ότι δυσκολευόμαστε με οποιαδήποτε πρόταση που μπορούσε ενδεχομένω να συνεπάγεται χαμελότερη προστασία καταναλωτών από τις στι εγχώριες αγορές Συχνά σε περίπτωση εναρμόνισης ε, μιλάμε για ελάχιστη ε, εναρμόνιση. Κατά περίπτωση, γιατί σε κάποιε περιπτώσει κοιτάμε και τι γίνεται κατά περίπτωση. Κοιτώντα λοιπόν τι γίνεται με το πακέτο τηλεπικοινωνιών, σε κάποια μέρη τη Ευρώπη οι καταναλωτέ. έχουν δικαιώματα τα οποία δεν έχουν οι καταναλωτέ σε άλλα τμήματα τη Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή πρότεινε. Η Επιτροπή μα ε, προτείνει ελάχιστη εναρμόνιση. Το Συμβούλιο ούτε καν αυτή την ελάχιστη εναρμόνιση δεν αποδέχεται. Μιλάτε για πλήρη εναρμόνιση λοιπόν, Επιτροπέ. Αν θα μπορούσατε να διαβάσετε ένα μήνυμα. Αν είναι να έχουμε εναρμόνιση, θέλουμε να υπάρχει κάτι που θα περάσει και το Συμβούλιο και να μην οδηγηθούμε σε υποβάθμιση προτύπων σε κάποιες χώρες. Η πλήρης εναρμόνιση δεν είναι η ίδια σε κάθε περίπτωση. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται ελάχιστη, σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται μέγιστη εναρμόνιση. Ο Επίτροπος. Ναι, αλλά επιτρέψτε μου να απαντήσω άμεσα. Όπως ξέρετε, αξιότιμη Πρόεδρε, συμφωνούμε. Συμφωνούμε στα θέματα αυτά. Οι απόψει τη Επιτροπή είναι ταυτόσιμε με αυτέ του Κοινοβουλίου στα θέματα αυτά. Να μην τα ρίξουμε όμω όλα στο Συμβούλιο σήμερα. Σίγουρα όμως υπάρχει πολύ, πολλά στοιχεία που μας αναστατώνουν. Αλλά ας μην ξεκινήσουμε εδώ σήμερα να τα λέμε. Um... Μάλιστα. Η Ρέτα, Thank you, Mr. Vice President. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε που ήρθατε και να μας μιλήσετε για την στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Ποια είναι τα σχέδιά σου γιατί είναι το geo-blocking σε ό,τι αφορά τα περιεχόμενα που έχουν αγοραστεί. Γνωρίζετε όμως το ότι το μεγαλύτερο τμήμα των έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διατίθεται προς πώληση διασυνοριακά. Δύο παραδείγματα να σας δώσω. Υπάρχουν πλατφόρμες όπως το YouTube που ήταν εικονικές για το πρόβλημα του geo-blocking και άλλες πλατφόρμες όπως η δημόσιοι σταθμοί εκπομπής που πάσχουν από το πρόβλημα αυτό. Και έτσι το να επιτρέψουμε την ε, διαβίβαση τέτοιων δεδομένων δεν θα βοηθήσει στο geo-blocking. Είσαστε διτεθειμένοι λοιπόν να προχωρήσετε μέχρι τέλους σε ό,τι αφορά το geo-blocking, τις γεωγραφικές αυτές ε, διαφορετικές μεταχειρήσεις. Ύστερα, το πρόγραμμά σας για το βάθμος. Και εδώ μία από τις ιδέες ε, για να βελτιωθεί η κατάσταση άμεσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί κατόφλε μιλάμε και υπάρχει όντως ε, αυτό προπτική. Να υπάρχει ένα ανατατό όριο, ένα κατόφλι μάλλον 130.000 ε, ευρώ ανακύκλω εργασιών και πόσο γρήγορα μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το όριο. Νίκολα. Ευχαριστούμε πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε που ήρθατε τώρα εδώ είμαστε τόσο συγκεκριμένα. Με μεγάλη μου ικανοποίηση άκουσα την εισήγησή σας και ένα από τα βασικά σημεία είναι αυτά για το μέλλον μας σε σχέση με την ψηφιακή ατζέντα. Δηλαδή, τι γίνεται, πώς θα έχουμε κάποια εφαρμογή της ψηφιακής οικονομίας για τον βιομηχανικό μας ιστό. Εγώ νομίζω ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί στον κόσμο με, ε, τις νέες τεχνολογίες στους νέους τομείς τη τεχνολογία. Ε, είμαστε όμω μεγάλο βιομηχανικό παραγωγό, οπότε νομίζω ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί πάρα πολύ να βοηθήσει όσον αφορά αυτόν τον στρατηγικό κλάδο και από πλευρά επίση ε, απασχόληση. Αυτό πάνω από τη βιομηχανία. Εγώ νομίζω ότι όπω εσεί αφήσατε να ενθεί από την παρέμβασή σα, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να επενδύσει πάνω σε αυτό. Οπότε γι' αυτό και εγώ θα ήθελα να μου πείτε ε, πιο συγκεκριμένα τι γίνεται, ποιες δράσεις πρόκειται να αναλάβετε ε, όχι μόνο για να υποστηρίξετε τη νέα ψηφιακή θεματολογία αλλά επίσης ε, ούτως ώστε η βιομηχανία να αποκτήσει νέες παραγωγές δυνατότητες καινοτόμες και βέβαια δυνατότητες συμβατές με τη νέα τεχνολογία τι γίνεται επίσης με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τι γίνεται με την ε, κλασική, την καθιερωμένη παραδοσιακή βιομηχανία, πώς είναι δυνατόν να έχουμε αυτό το μετασχηματισμό προς ε, την, καινούρια την ψηφιακή ε, παραγωγή, κατασκευή, μεταποίηση, γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική. Και να δούμε πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι νέες ιδέες ακόμα και στους προδιασιακού τομείς της οικονομίας και της βιομηχανίας. Και άλλα θα σας πω, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να τοποθετηθούν όλοι οι συνάδελφοι. Thank you, Chair, and thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο σε αυτά που είπε η Ιουλία σε σχέση με την κινητικότητα του ψηφιακού περιεχομένου και το γεωγραφικό αποκλεισμό, το geo ακούσαμε και είναι θετικό. Θέλετε να δράσετε στον τομέα αυτό, να δεν μα δώσετε λεπτομέρειες. Αυτό είναι το κέριο σημείο. Με ποιο τρόπο θα μπορούμε να προχωρήσουμε με, σε κάποια μορφή ε, δυνατότητας μεταφορών των δικαιωμάτων αυτών χωρί να δημιουργηθεί κάποια ευρωπαϊκού χαρακτήρα αδειοδότηση. Θα ήθελα λοιπόν να μου δώσετε περισσότερε πληροφορίε, Ξέρω ότι αυτά θα γίνουν δημόσια σε λίγε εβδομάδε, αλλά ό,τι και να μου πείτε θα είναι πολύ θετικό. Επίση, ένα θέμα πιο γενικό ο λεγόμενος ελέφαν, ελέφας ενδοματίο. Αν θέλουμε να είναι πράγματι επιτυχημένη η ψηφιακή μας αγορά, θα πρέπει να αλλάξει τα τωρινά επιχειρηματικά μοντέλα. Δεν μπορεί να το πετύχουν αυτό χωρίς να τα ανατρέψουν. Για παράδειγμα, η Uber, MBMB, Google, όλες αυτές οι εταιρείες σε ψηφιακό επίπεδο είναι πάρα πολύ επιτυχημένες και σε επίπεδο καταναλωτών είναι επιχειρηματικά επιτυχημένες αλλά έχουν ανατρέψει τα προηγούμενα μοντέλα και η απάντησή μας ήταν κάπως ιδιαίτερα μονοκόμματη γιατί τα μοντέλα μας δεν είναι για τον επιγραμμικό κόσμο, είναι για τον offline κόσμο, τον κόσμο εκτός διαδικτύου. Δύο ερωτήματα. Πρώτον, πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε τους επιχειρηματίες του διαδικτύου και να τους κάνουμε παγκόσμιους πρωταθλητές στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν κάθε φορά που κάνουν κάτι που είναι επιτυχημένο τους βάζουμε κανονισμούς που τους καταστρέφουν το μοντέλο τους. Και δεύτερον, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να πάρουμε ε, κατευθύνσεις από άλλους νομοθέτες στα κράτη-μέλη. Θεωρείται ότι υπάρχει μια κατανόηση μεταξύ των εθνικών νομοθετών και των ευρωπαίων νομοθετών ότι θα πρέπει να αλλάξουμε πολλούς από τους κανονισμούς μας για να μπούμε πλήρως στον ψηφιακό χώρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε και εγώ κατανοώ το γεγονός ότι πάντα σας ενδιαφέρει να βελτιώσουμε πάντα το θέμα των πωλήσεων στο διαδίκτυο, να μειώσετε τα εμπόδια για διαμεθοριακές πωλήσει. Αλλά αυτό συνδέεται και με την τωρινή δομή του ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε σαν σχέδιο να ξεκινήσετε κάποιες αλλαγές για το σύστημα φορολογίας ΦΠΑ που αποτελεί πράγματι και ένα εμπόδιο για διαμεθοριακές πωλήσει δεύτερον. Και αυτό έχει να κάνει με την θέση των πρωτοπόρων ψηφιακών εταιριών στις χώρες μας. Υπάρχουν οι λεγόμενοι ηγέτες σε ψηφιακό επίπεδο σε κάθε χώρα και που είναι σε ισχυρή θέση για να μπορέσουν να μεταλαμβαδεύσουν τις ιδέες της ψηφιακής αγοράς. Θα χρησιμοποιήσετε λοιπόν αυτούς τους ηγέτες με κάποιο τρόπο ή όχι. Με ποιο τρόπο κιόλας θα το κάνετε. Η κυρία Μακλάρκιν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι όλοι μας θέλουμε να δούμε μια πλήρως λειτουργούσα ψηφιακή εσωτερική αγορά, να δώσουμε μια περαιτέρω όθηση για να έχουμε περισσότερη ανάπτυξη και θέσεις απασχόληση. Θα ήθελα και η ομάδα μου θα ήθελε να γίνει αυτό επί τη βάση πραγματικών στοιχείων και αποδείξεων. Έχουμε κάνει λοιπόν διαβουλεύσεις, έχουμε κάνει μελέτες αντικτύπου, καταλαβαίνουμε ότι οι πρωτοβουλίε οι οποίες προτείνονται ή εξετάζονται ή ερευνούμε βασίζονται σε αυτό το στόχο. Όταν πρόκειται λοιπόν για το γεωγραφικό αποκλεισμό, τον μη δικαιολογημένο γεωγραφικό αποκλεισμό, θα ήθελα να ξέρω η Κομισιόν έχει κάποια στοιχεία που να δείχνουν ότι θα υπήρχε πραγματικά κάποια όθηση για ανάπτυξη <clears throat> εάν η ευδοκιμούσε αυτή η πρωτοβουλία για την άρση του γεωγραφικού αποκλεισμού. Επίσης ζούμε σε έναν κόσμο που προσπαθούμε όλοι να τον πλησιάσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτόν τον κόσμο, τον ψηφιακό κόσμο. Και ο χρόνος που ξεκινάμε τις δράσεις σε σχέση με τη χρονική στιγμή που η αγορά αρχίζει να ξεκινάει, είναι τέτοια χρονική στιγμή που είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει κανείς να καταλάβει τι γίνεται. Παραδείγματος χάρη με την εξόριξη δεδομένων, η εξόριξη κειμένου, αυτά είναι πράγματα τα οποία οι ο οικονομικός κλάδος προσπαθεί να βρει ένα μοντέλο το οποίο είναι βιώσιμο με αδειοδότηση κτλ. για να λειτουργήσει αυτό. Αν σε αυτό το πολύ πρώιμο στάδιο εμείς προτείνουμε νομοθεσία μπορεί να τροχοπεδίσουμε την ανάπτυξη αυτών των αγορών, να επιτρέψουμε να στρεβλωθούν με την παρέμβασή μας λοιπόν σε πρόωρο στάδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε προβλήματα. Θέλω όμως να συγχαρώ την Κομισιόν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ότι καταλαβαίνει ότι θέλει να υποστηρίξει τον δημιουργικό τομέα για να τους προστατεύσει από παραδιάσει των δικαιωμάτων τους με μια στεναρή διαδικασία συνόμευσης και εφαρμογής. Πρέπει να πολύ προσεκτικοί όταν λέμε ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα σταθερό πλαίσιο για την εφαρμογή των ε, δικαιωμάτων των καλλιτεχνικών δημιουργών. Δεν τους ε, περιορίσουμε συγχρόνως με το να περιορίσουμε τη χρήση αυτών των δικαιωμάτων μη τους δίνοντας τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν αυτά τα δικαιώματα και σε άλλους χώρους. Γιατί αυτά τα οποία θα πετύχουν από τη διαδικασία για παράβαση των δικαιωμάτων τους δεν θα είναι επαρκή και θα συνεχίσει να υπάρχει αυτός ο κύκλος ο οποίος θα είναι αρνητικός για Πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να είναι δημιουργική, με το να αποκομίσουν την αξία την οποία πρέπει να πάρουν από τα δημιουργήματά τους. Αν θέλετε να απαντήσετε, λέει πρόεδρο, σα ευχαριστώ και πάλι. Σα ευχαριστώ για τι ερωτήσει σα. Ρωτήσατε για το γεωγραφικό αποκλεισμό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ότι το να επιτρέψουμε μόνο να μεταφέρετε το περιεχόμενο δεν αποτελεί λύση. Θα πρέπει να επιτρέπουμε και πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό. Όπως όλοι ξέρουμε, η σημερινή κατάσταση είναι μια κατάσταση η οποία είναι αμοιβαία δεν είναι προς όφελος θα θέλαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια κατάσταση αμοιβαία επωφελή. Θέλω να πληρώσω, θέλω να έχω ένα περιεχόμενο και οι δημιουργοί θα έχουν πιο πολλά χρήματα για να δημιουργήσουν πιο, πολλά, α, πολλές ταινίες. Έτσι όλοι θα είναι κερδισμένοι. Και ε, αυτό είναι ο σκοπός μου. Σήμερα 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι περίπου θα ήθελα να έχουν διασυνοριακή πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο, σε μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία από κάποια άλλη χώρα της Ένωσης. Δεν μπορούν όμως. 271 271 ε, εκατομμύρια ε, ταξίδια γίνονται για να έχει ο κόσμος πρόσβαση σε τέτοια περιεχόμενα. Για να έχει ο κόσμος πρόσβαση σε τέτοια περιεχόμενα, αλλά κατά κανόνα δεν μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό που θέλει. Τους μπλοκάρει. Και δεν μιλάω για κάποιες μικρές ε, μειοψηφίες όταν μιλώ για την κατάργηση του γεωγραφικού αποκλεισμού, αλλά δεν θέλω και να καταστρέψω και την αρχή της ε, εδαφικότητας στην αξιοποίηση των ε, προϊόντων αυτών. Ξέρω ότι προτείνεται πανευρωπαϊκές άδειε, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις όταν είναι μικρή η παραγωγή ποιοι είναι δεσμένοι να αγοράσει αυτές τις αγορές. Κανείς δεν θέλει να αγοράσει πανευρωπαϊκές ε, άδειες όταν είναι μικρός παραγωγιός. Ούτε θέλω ένα σύστημα release Windows. Ξέρω ότι υπήρχαν άτομα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι αυτή την Επιτροπή, αλλά στην προηγούμενη, που ήθελε να αλλάξει αυτό το σύστημα. Αλλά με την ψηφιακή ενιαία αγορά δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτό το σύστημα. Καταρχά ε, ε, για τι ταινίε στο σινεμά, DVD, video on demand. Εδώ θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω πρόσβαση διασυνοριακή σε αυτά τα περιεχόμενα. Πολλά από αυτά τα άτομα που υποτίθεται ότι προστατεύουν τους δημιουργούς δεν ε, προσέχω τελικά ποια είναι η πραγματικότητα. Και έχω πει ήδη στην ακρόαση μου στο Κοινοβούλιο ότι σε ένα άρθρο του, του Twitter Link έλεγε ότι 29% των Καναδών ε, βλέπουν ταινίες ε, στο Netflix με αμερικανικές διευθύνσεις IP. και σύμφωνα με το άρθρο αυτό ένα τρίτο των Καναδών βλέπουν ταινίε μέσω του Netflix με VPN και μέσω αμερικανικών ε, διευθύνσεων IP. Και σύμφωνα με ένα άλλο άρθρο, δεν θυμάμαι την πηγή, Δεν θυμάμαι το άρθρο, αλλά είναι δύσκολο πάντα γιατί πηγαίνουμε μέσω συνδέσμων από ένα άρθρο στο άλλο. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο αυτό, 13 εκατομμύρια άτομα στην Κίνα χρησιμοποιούν το VPN και βλέπουν ταινίες τέτοιες. Ξέρουμε λοιπόν πόσο εύκολο είναι μέσω χρήσης VPN να έχει κανείς πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο. Άρα ουσιαστικά στην πραγματική ζωή ο γεωγραφικός αποκλεισμός δεν αποτελεί πρόβλημα τεχνικός πόσο. Είμαι όμως απόλυτα βέβαιος ότι ο κόσμος θέλει να είναι έντιμος θέλει να καταναλώνει με ειλικρινή τρόπο και να πληρώνει για αυτό που καταναλώνει. Σήμερα όμω δεν δεχόμαστε τα χρήματά του ουσιαστικά. Ένα παράδειγμα να σα δώσω για το Spotify και την εμπειρία τη Αυστραλία. Όταν η το νόμιμο κατέβασμα του Spotify αυξήθηκε, μειώνονταν τα παράνομα κατεβάσματα από torrent. Είχε λοιπόν μια αναλογία μεταξύ παράνομου και νόμιμου κατεβάσματο. Όλοι ξέρουμε ότι η πειρατεία δεν ε, κοστίζει τίποτα. Αν οι παροχοί όμω υπηρεσιών μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες καλύτερη ποιότητα, ψηλότερης ταχύτητα. ο κόσμος ε, θέλει να πληρώσει. Και πάλι θα ήθελα να επαναλάβω ότι εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω του δημιουργού θα ήθελα να του δώσω πιο πολλά χρήματα. Γιατί θέλω πραγματικά, στόχος μου είναι να υπάρχει ανταμοιβή των δημιουργών. Πρέπει λοιπόν να δούμε και το θέμα της εφαρμογή του νόμου, όπως αναφέρεται. Θα ακολουθήσουμε την αρχή follow the money. Κάποιε επιχειρήσει επιχειρήσεις χρηματοδοτούν τις πλατφόρμες αυτές, αυτές τις εφαρμογές που επιτρέπουν είναι το παράνομο κατέβασμα ψηφιακού περιεχομένου. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και αυτούς τους φορείς. Επαναλαμβάνω, στόχος μου είναι να δημιουργηθεί μια αμοιβαία αποφελή κατάσταση. Στόχο μου είναι να προστατευτεί τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία. αλλά να υπάρχει και διασυνοριακή πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο και να υπάρχει πρόσβαση του κόσμου στα περιεχόμενα αυτά, γιατί πραγματικά το αξίζουν. Κάτι άλλο τώρα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να επαναλάβουμε την πρόταση αυτή που έγινε το 2004 μέχρι το 2008, ήδη από τότε, να υπάρχει ένα αρκετά υψηλό κατόφλι. Εγώ προτείνω να είναι τα 100.000 ευρώ αυτό το όριο. Ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ήδη υπάρχει ένα υψηλό κατόφλι, 81.000 ε, λίρες Αγγλίας, ε, οι επιχειρηματίες ε, διαμαρτύρονται για την υψηλή γραφειοκρατία. Θα πρέπει να ακούσουμε, να εισακούσουμε αυτές τις διαμαρτυρίες. Η πρόταση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ξέρετε, ε, απορρίφθηκε από τα κράτη-μέλη. Ελπίζω αυτή τη φορά τα κράτη-μέλη να πάρουν πιο στα σοβαρά αυτή την πρόταση. Για το κλάδο τώρα και την τυποποίηση. Να μιλήσω και πάλι για θέματα τυποποίησης και διαλειτουργικότητας. Mm. Τα εργαλεία αυτά σε κάθε περίπτωση θα βοηθήσουν τον κλάδο να περάσει την ψηφιακή φάση. Όπως θυμάστε, η εποχή του GSM ήταν πραγματικά έντοξη εποχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα όμως ε, πολύ λυπάμαι που σας ε, λέω ότι σε ό,τι αφορά το 4G έχουμε μείνει πίσω. Δεν έχει γίνει αυτό πραγματικότητα ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες. Και λίγαν συντόμως θα πρέπει να υπάρξουν νέα πρότυπα για το 5G και πραγματικά ελπίζω να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε τη διαδικασία τυποποίησης με τις προτάσεις αυτές με μια διαδικασία πιο δύσκολη από ότι αυτή του Φρέζη και του Φόρτζη. Πρέπει να μιλήσουμε πολύ πιο πολύ για τα δεδομένα όταν μιλάμε για την οικονομία των δεδομένων. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για την κατοχή των δεδομένων, την διακτησία των δεδομένων. Όταν μιλάμε για δεδομένα και για προστασία, μιλάμε μάλλον κυρίως για προστασία δεδομένων. Θα πρέπει όμως να συζητήσουμε και το θέμα των δεδομένων ως μια, ένα φυσικό πόρο, ένα αγαθό πολύτιμο. Για τις νεοφυείς τώρα. Οι νεοφυείς όντως δημιουργούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα πιο ευέλικτα άτομα ουσιαστικά. Με ταχύτατες αντιδράσεις σε όλες τις ευκαιρίες, όλων των ειδών τις ευκαιρία. Θα πρέπει το πλαίσιο, το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι φιλικό προς τις νέες συσταθεί εταιρείε. Γιατί να χρειάζεται να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάνε στη ΣΥΠΑ οι νεοφύης για να αναπτυχθούν. Γιατί δεν μπορούμε να καθίσουμε τις έξυπνες ιδέες τα ευθεία, στα μυαλά στην Ένωση. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κλίμα πιο φιλικό στις νεοφύης εταιρείε. Και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των νεοφιών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποφεληθούν πιο πολύ από κάθε άλλο κλάδο από την ε, ψηφιακή ένωση. Όταν όμως δημιουργούμε την ψηφιακή αυτή ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το κάνουμε για λίγους, δεν το κάνουμε για τους εκλεκτούς, το κάνουμε για όλους, για τις επιχειρήσεις μα. αλλά και για επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες. Για την ε, μεταφερσιμότητα. Δεν θέλω να καταστρέψω ή να παραβιάσω αυτή την αρχή της εδαφικότητας. Αλλά δεν θέλω να έχω απόλυτη προστασία της εδαφικής αποκλειστικότητας. Αν συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο, τότε η δυνατότητα μεταφοράς των ε, περιεχομένων του ψηφιακού περιεχομένου, δεν θα έχει κανένα νόημα. Θα πρέπει και πάλι να επιτρέψουμε διαμεθοριακή πρόσβαση και δυνατότητα μεταφοράς του ψηφιακού περιεχομένου προς όφελος των πολιτών μας. Ξέρω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να αλλάξουν το σύστημα των κανονισμών Του βεβαίω θα το κάνουν. Και υπάρχουν αποχρόντες λόγοι για να μπορέσουν να τροποποιηθούν αυτοί οι κανονισμοί. Το ξέρετε καλύτερα εμού βάσει αναλύσεων που έχουν εκπονηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τιμή της μη Ευρώπης σε ψηφιακό επίπεδο είναι πολύ ψηλή. 340 δισεκατομμύρια μη ευρώ θα είναι το κόστος της μη ψηφιακής Ευρώπης. Και δεν μιλάω για χρήματα μονάχα. Μιλάω και για θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρώπη. Το να υπάρχουν διακρίσεις μέσω του γεωγραφικού αποκλεισμού εναντίον ορισμένων πολιτών μέσα στον 21ο αιώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι παραδεκτό. για το σύστημα ΦΠΑ και για το τι προβλέπουμε για να αλλάξουμε αυτό το σύστημα. Για όλα τα θέματα φορολογικού χαρακτήρα είναι ο Επίτροπος Μοσκοβισή ο οποίος θα ασχοληθεί. Και ξέρετε ότι όλοι οι Επίτροποι συνεργάζονται με μεταξύ τους, αλλά έχουμε αποφασίσει ότι όταν, προ... όταν μιλάμε για δεξιότητες θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια ολιστική προσέγγιση και δεν θα διαχωρίσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες από τις μη ψηφιακές δεξιότητες. Αλλά θα τα αντιμετωπίσουμε από κοινού. Η πρόθεσή μας είναι λοιπόν να συνεχίσουμε σε συνεργασία με, την, ε, ε, με τους λεγόμενους ψηφιακούς πρωταθλητές ε, θα συνεχίσουμε αυτήν την συνεργασία και το είχα κάνει και στη δική μου ε, διάρκεια της δικής μου, δικής μου εντολής και όταν επισκεπτόμουν κράτη-μέλη πάντα προσπαθούσα να έρθω σε επαφή με τους ψηφιακούς πρωταθλητές στα κράτη αυτά μέλη. Για τις εκθέσεις που τη δημόσια διαβούλευση, όλα αυτά είναι απαραίτητα. καθήμενος δίπλα στην κυρία Πρόεδρο, η οποία ενδιαφέρεται για την προστασία των καταναλωτών και για την καλύτερη ρύθμιση στην εσωτερική αγορά, δεν μπορώ να τρέφω ούτε καν αμφιβολίες σε σχέση με την ισχύ αυτών των αρχών. Δεν φαντάζομαι ότι θα μπορούσα να είχα μια διαφορετική άποψη σε σχέση με τις δημόσιες διαβουλεύσεις και την ε, έκθεση αντικτύπου. για την εξόριξη δεδομένων και κειμένων. Είναι διαφορετική κατάσταση σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι επιστήμονες έχουν πρόσβαση σε αυτά τα καινοτόμα εργαλεία. Αυτοί οι οποίοι εργάζονται με μαζικά δεδομένα, με μεγάλες ποσότητες δεδομένων, χρησιμοποιούν την εξόριξη δεδομένων και οι επιστήμονες σε άλλα κρατημέλη λυπάμαι εδώ που το λέω δεν το κάνουν. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι επιστήμονές μας σε υψηλό επίπεδο πάντα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε μεγάλα σύνολα δεδομένων διότι όπως ξέρουμε είναι δυνατόν να βρει κανείς κάθε είδους συσχετισμούς από τα μεγάλα αυτά δεδομένα που θα εξετάσει κανείς. Μπορεί να βρει συσχετισμούς λοιπόν και σχέσεις χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα και να μπορέσει να κερδίσει ιδέες για θετικές απαντήσεις από την εξόριξη στοιχείων και κειμένου. Νομίζω λοιπόν ότι έχω δώσει μια απάντηση σε όλα τα ερωτήματά σας. Έχω μάλλον τέσσερις αγωνιτές, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία και Rosa and I'm αλλά επειδή πρέπει να φύγω, δεν μπορώ ψηφιακά να πάω, πρέπει σωματικά υλικά να μεταβώ στην πατρίδα μου. Απλώς να σα πω ότι πολλές φορές έχουμε κάποιες ε, τρομερές επιτυχίες στην Ευρώπη όπως έγινε αυτό πρόσφατα γιατί έχουμε έξι από τις δέκα ε, κορυφαίε ε, οικονομίες που ψηφιακά συνδεδεμένε βρίσκονται στην Ευρώπη. Οι δύο από αυτές βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Τα συζητήσαμε επίσης αυτά ήδη και έχουμε αυτές τις εταιρείε μονόκερους που μιλούμε ότι αξίζουν δις. Είναι 30 στην Ευρώπη, 99 στην ε, Αμερική ε, και την περασμένη εβδομάδα δε. Είχαμε και έναν επιχειρηματία στην τεχνολογία ηλικίας 62 που βρήκε ένα μικροκύκλωμα, το εφήβρε, σε σχέση με τα φορητά τηλέφωνα που άμα χαθούν ε, κάτι ε, εκπέμπουν κλπ. Οπότε είναι τώρα ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής μικρο, ε, μικροκυκλωμάτων. Να, βλέπετε τι γίνεται εδώ. Για το crowdfunding επίσης είμαστε ε, πρωτοπόροι. Στη, στα TechFin επίσης είμαστε πολύ πιο μπροστά από ό,τι είπα. Κάποιοι γκρινιάζουν και λένε ότι δεν αποδίδουμε, αλλά όχι, είμαστε προθαλητές. Ας εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε περισσότερες από αυτές. Κάθριν Στάιλ. Δίκη, σε ευχαριστώ. Αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα ο κόσμος. Ε, ένα στους δύο ανθρώπους τώρα έχουν ε, smartphone, έχουν ε, λογαριασμό στην τράπεζα. Είδατε πόσο τους φτάνει, πόσο γρήγορα τους αγγίζει τεχνολογία. Είδατε τι γίνεται με την ψηφιακή στρατηγική που μας παρουσιάσετε. Τώρα, πες μας κάτι για τα μαζικά δεδομένα. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήδη κινείται σε αυτό το πλαίσιο γιατί έχει τις υποδομές τι μπορεί να γίνει παραπέρα και για το copyright ποιες μπορεί να είναι οι ρεαλιστικές μας προσδοκίες για μεταρρύθμιση πρώτη υποποίηση μας είπατε και για την διαλειτουργικότητα για ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις ε, συμβάσεις διαγωνισμούς προμηθειών θα πρέπει όμως τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν περισσότερο μεταξύ τους. Ακούσαμε και για τις δεξιότητες, μας είπατε για την ε, Επίτροπο Τάισεν, με τι ασχολείται. Επομένω πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Και οι καθηγητές τους υπολογιστές στην Βρετανία είναι μόνο 7% γυναίκες. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να έχουμε περισσότερες γυναίκες που να κάνουν σταδιοδρομία στην πληροφορική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάντως, για να ολοκληρώσω, περιμένω ανυπόμονα την πρότασή σας θα δημοσιοποιηθεί στις 6 Μαΐου. we have very ότι έχουμε γυναίκες με προσωπικότητα εδώ στην Επιτροπή. Η Εύα. Βίκη, σε ευχαριστώ. Εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι ισορροπημένα σήμερα. Γιατί είχαμε τη στον κύριο Τράπεζα στη Σόφη με τον ε, κύριο Επίτροπο και ήρθαν ε, ε, ο Πρωθυπουργό, οι Υπουργοί. Πολλοί Υπουργοί. Όμω τότε εγώ ήμουν η μόνη γυναίκα. Να και αυτό τώρα σκεφτόμουν. Πόσε τέτοιες ε, συζητήσεις οργανώνουμε εδώ. Όχι, όχι, τα πράγματα είναι ισορροπημένα. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε που ήρθατε. Σας ευχαριστώ όμω και που ταξιδέψατε και μέχρι τη Σόφια. Μας υποσχεθήκατε ότι θα συνεργαστείτε στενά με το Κοινοβούλιο και θα έρχεστε εδώ τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψει. Κατά εκείνη λοιπόν την διάσκεψη τη συνάντηση με μερικές μέρες είχαμε Επιτροπή Κοινοβούλιο και τι εθνικέ αρχέ, την κυβέρνηση. Και είπαμε ότι για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ε, ψηφιακή αγορά χρειάζεται μια ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεσματική, φιλική στο χρήστη κλπ. Για να ρωτήσω κάτι που δεν το έχει ρωτήσει κανείς μέχρι τώρα. Πρώτον, για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες. Θέλουμε επιχειρηματίες αλλά και οι Ευρωπαίοι να μπορούν πλήρω να ωφεληθούν από τις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κλπ. Και έτσι να ανέβουν οι δεξιότητες τους ηλεκτρονικές. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνεται, λέω μέσω της επαγγελματική κατάρτισης και μέσω της παιδείας. Να, που η ψηφιακή στατική μπορεί να βοηθήσει. Η ψηφιακή νέα αγορά. Χρειάζεται τώρα ε, και εργοδότες και εργαζόμενοι με υψηλή κατάρτιση. Οπότε αυτή η νέα ε, στρατηγική που θα μας την παρουσιάσετε στις 6 Πέμπτου, με τι εργαλεία πρόκειται να βοηθήσει τις ηλεκτρονικές δεξιότητες, από μια τρυφερή ηλικία. Τι είναι με τις ε, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, πώς θα λειτουργήσουν, πώς ξέρετε, ε, πρόκειται να βοηθήσουν την εμπιστοσύνη επιχειρήσεων και πολιτών για τις ηλεκτρονικές, τις ψηφιακές μάλλον υπηρεσίες. Η δε παροχή, η προσφορά τέτοιων δημοσίων υπηρεσιών δεν θα φέρει προς αξία εάν δεν υπάρξει εμπιστοσύνη από τους πολίτες γιατί δεν θα χρησιμοποιήσουν τεχνολογία. κυριαλογική θα μπορούσε να ισχύει και για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οπότε, η νέα στρατηγική για την ψηφιακή αγορά τι λύσεις θα δώσει. Θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη των πολιτών. Γιατί αυτά έρχονται και με ρωτάνε καθημερινά οι καταναλωτές. Κύριε Σαλτεμόζα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω δανέζικα. Commissioner, thank you for, uh, coming here uh, and, I am really, really, really... Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και πραγματικά προσβλέπω να δω την παρουσίαση των προτάσεων, των συστάσεων αναχώρα. Αγγλικά μίλησα τελικά. <laughs> Now I will speak ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας λοιπόν. Χάρηκα ιδιαίτερα που ήσασταν εδώ μαζί, μα μαζί μας και για τις συγκεκριμένες προτάσεις που κάνατε. Νομίζω ότι πολλά μας βρίσκουν σύμφωνου σε ό,τι αφορά τις γενικότερες αρχές που προτείνατε για την ε, ψηφιακή ενιαία αγορά. Αλλά, όπως ξέρουμε, ο διάολος κλείβεται στις λεπτομέρειες. Και πριν θέσω τις ερωτήσεις μου, θα ήθελα να πω το εξή το θέμα του γεωγραφικού αποκλεισμού και της φορητότητας φυσικά συμφωνώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Αλλά μία ερώτηση συγκεκριμένη θέλω να σας κάνω. Έχετε σκεφτεί ποιες θα μπορούσαν οι συνέπειες για την ε, πολιτισμική ποικιλία στην Ευρώπη, τη γλωσσική ποικιλία, την πολιτισμική ποικιλία. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Ένα παράδειγμα το οποίο συχνά ακούμε για το Netflix, για παράδειγμα. Ναι, καλό και είναι φυσικά δεδομένο ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το VPN, το VPN αλλά ίσως να αντιμετωπίσουμε πολιτισμικές και γλωσσικές προκλήσεις. Αν οι νέοι τα παρακολουθούν αυτά χωρίς ε, πρόβλημα, αλλά ε, αντιμετωπίσουν προβλήματα οι πιο ηλικιωμένοι. Έχετε λοιπόν αναλογιστεί τις συνέπειες για την πολιτισμική επικλεμορφία. Είναι όλα θετικά και θα πρέπει να επικεντρωθούμε όμως και στις συνέπειες τις πολιτιστικές και μήπως θα έπρεπε να πάρουμε μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την ε, μορφή αυτή. Ευχαριστώ πολύ, η επόμενη μιλήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους μας ότι πραγματικά κάνετε αυτά που λέτε. Είχατε υποσχεθεί ότι θα συνεργαστείτε στενά μαζί μας και το κάνατε Χαιρόμαστε που έρχεστε τόσο δακτικά λοιπόν εδώ στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα. Να κάνω κάποιε ερωτήσεις τώρα σε ό,τι αφορά την επερχόμενη στρατηγική για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Η πρόταση, είπατε, θα ανακοινωθεί, αλλά θα ήθελα να ξέρω ποιο νομικό εργαλείο θα προτιμούσατε. Κανονισμό ή οδηγία θα προτιμούσατε. Επίσης, σε διάφορες περιπτώσεις ε, αναφερθήκατε ότι χρειάζονται ένα τολμηρό όραμα. Αυτό μας λέει οι επιχειρήσεις τουλάχιστον. Θα προτείνετε νομοθετική δράση για να διασφαλίσετε υψηλής ποιότητας ε, διασυνοριακές υπηρεσίες σε λογική τιμή, γιατί από ό,τι ξέρετε η αγορά είναι καταγραμματισμένη σε 28 εγχώρες αγορές, οι οποίες έχουν ε, κυρίαρχη θέση σε κάθε χώρα και δεν είναι πάντα τόσο ανοιχτές, δεν είναι τόσο καινοτομικές. Ε, δεν είναι οι πιο αποδοτικές αν θέλετε πάντα. Θέλετε να δημιουργηθούν πιο καινοτόμες λύσεις καινοτομίας. Σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο πελάτης του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν χρειάζεται πάντα παράδοση στο σπίτι του πέντε φορές την εβδομάδα από τις 9 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Όπως ξέρετε υπάρχουν πολύ πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί τρόποι ε, παράδοσης. Όπως ξέρετε παράδοση σε βενζινάδικα, σε λόκερ, σε διάφορες τοποθεσίες. Ερευνάτε λοιπόν ε, ποιες είναι αυτές οι λύσεις, οι πιο αποτελεσματικές λύσεις, οι νέες λύσεις για τις καινοτομικές υπηρεσίες. Είχαμε μια εξαιρετική παρουσίαση της ανάπτυξης ODR για την πλατφόρμα αυτή και πώς εξελίσσεται. Ήταν πολύ ωφέλιμη. Ελπίζουμε να είναι αυτή η πλατφόρμα έτοιμη στα, στις αρχές του επόμενου έτους και ελπίζουμε να υπάρξει και εντομία σε όλη την αγορά με την ταχύτητα Επίσης, να πω δύο λόγια για την ε, οικονομία για την κοινή αυτή η οικονομία. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι αν ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναλάβουμε τα ενία, την ηγεσία, τα κρατη πολύ απλά θα καταγερματίσουν το νομικό πλαίσιο, δημιουργώντας ένα τοπίο εντελώς διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών. Και εδώ, πολύ σπανίως σήμερα διαπιστώνουμε ότι οι εταιρείε απευθύνονται σε εμάς τα ευρώ από όργανα. Αυτό σχεδόν ποτέ δεν συμβαίνει. Ποτέ δεν μας ζητούν να ρυθμίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προγραμματίζει δράσεις, ε, ναι, να λάβει δράση και σε ό,τι αφορά τις 6 Μαΐου. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και στην ομάδα εργασία μας την προηγούμενη εβδομάδα. Ακούσατε ποιε ήταν η ανησυχία των εμπλεκόμενων φορέων υπάρχουν πολλά καινοτόμα άτομα και επιχειρήσει, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, που φεύγουν, πάνε στη ΣΥΠΑ. Γιατί εκεί μπορούν να αναπτυχθούν καλύτερα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Αναφερθήκατε στον κατακαιρματισμό, αλλά πραγματικά θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό. Και συμφωνώ με αυτή την συνολική προσέγγιση στο θέμα. Αυτό το ληστικός, ε, συνολικός είναι πολύ μοντέρνα έκφραση. Αλλά αν τη θέλουμε αυτή την προσέγγιση, τη συνολική την ολιστική, πιστεύω ότι η στρατηγική για την ενιαία αγορά θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ενιαία αγορά για τις τηλεπικοινωνίες. Γιατί το, η περιαγωγή, η περιαγωγή δεδομένων είναι τμήμα των τηλεπικοινωνιών και της σχετικής ενιαίας αγοράς και θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται. Τέλος, αυτό το λέω ως πρόεδρος της ομάδας εργασίας για την ψηφιακή ενιαία αγορά και να ευχαριστήσω και όσους συμμετέχουν τόσο ενεργά στις συναντήσεις μας. Θα ήθελα να οργανώσω συγκεκριμένες ε, συζητήσεις με τις υπηρεσίες σας, γιατί οι βουλευτές ε, το ζητούν μετά την έγκριση από το Σώμα των Επιτρόπων της ενιαίας ψηφιακής στρατηγικής θα μπορούσατε να μας ε, πείτε ποιοι είναι οι αρμόδιοι διευθυντές από τη Γενική Διεύθυνση για να συζητήσουμε κατά περίπτωση με τους αρμόδιους τα σχετικά κεφάλαια, τα τμήματα της στρατηγικής. Μάλλον 12-13 Μαΐου θα διοργανωθεί η επόμενη συνεδρίαση. Βλέπω λοιπόν τη δέσμευσή σας, βλέπω και πόσο εντατικά δουλεύουν οι υπηρεσίες σας. Είμαι βέβαιη λοιπόν ότι θα συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία, θα έχουμε μεγάλο όγκο δουλειά, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και μόνο έτσι έχουμε πραγματικά την ευκαιρία να επιλεάσουμε την ψηφιακή αγορά της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Στενή συνεργασία λοιπόν, όχι με σας μόνο προσωπικά, αλλά και με τις υπηρεσίες σας. και θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση από κοινού στο Συμβούλιο προκειμένου τα κρατημέλη να μα μπλοκάρουν σε ό,τι αφορά την πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ε, ερώτηση για τις ηλεκτρονικές προμήθειες και το θέμα της διαλειτουργικότητας. Όπως ξέρουμε όλοι, οι ηλεκτρονικές προμήθειες είναι ιδιαίτερα εξελιγμένες στην Πορτογαλία. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, όταν μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις ηλεκτρονικές προμήθειες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται να εξοικονομήσουμε 50 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πάρα πολλά λεφτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες μας, εν γέννη, θα αποκομίσουν κάποιο όφελος από όλα αυτά. Κάποιες εταιρείες τώρα θα χάσουν. γιατί οι αγορές τους δεν θα είναι πια τόσο προστατευμένες. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το στόχο της ενιαίας αγοράς της απουσίας συνόρων και δεν είναι προστατευτικός ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξω τις ηλεκτρονικές προμήθειες και να υποστηρίξουμε λοιπόν όλες τις καινοτόμες ε, λύσεις στον τομέα αυτό που μπορούν να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γυναίκες στην πληροφορική. Είναι πρόβλημα αυτό. Μόνο 20% από τα άτομα που εργάζονται στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών είναι γυναίκες. Αλλά έχουμε διαφορετικές παραδόσεις, ιστορικές κτλ. Τι παραδόσεις μπορούμε να επικαλεστούμε όταν μιλάμε για πληροφορική, για υπολογιστές. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικές γενιές. Δεν είναι πατροπαράδοτες μορφές παραδόσεων από το μεσαίωνα. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε πολύ σοβαρά για τα θέματα αυτά και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι και οι γυναίκες μπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά στον τομέα αυτό από ότι και οι άντρες. Εντάξει. Εμπιστοσύνη. Α, για τις 6 Μαΐου πρώτα. Ναι, ναι, ναι, 6 Μαΐου. όπως ελέγχεται πολλές φορές. Ήδη πριν από τη συνεδρίασή μας αυτή, εμείς θα προτείνουμε μια στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά στις 6 Μαΐου. Για τις δεξιότητες, η Επίτροπος κυρία Τάισεν θα παρουσιάσει μια ολιστική στρατηγική για τις δεξιότητες και τις ικανότητες. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να βάλουμε και στο σχολικό πρόγραμμα των σχολείων μας την χρήση γλωσσών προγραμματισμού που δεν είναι και πολύ εύκολο. Όπως ξέρουμε, ο τομέας αυτός είναι ο τομέας ο οποίος παίζει μεγάλο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη. Δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1,8 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης, αλλά το 2018 σύμφωνα με τις προβλέψεις θα είναι 4,8 οι θέσεις εργασίας εκατομμύρια. Μόνο Μια τέτοια αύξηση λοιπόν κατά 3 εκατομμύρια, αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να τα προωθήσουμε. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτή την πρόκληση. Πολιτιστική πολυμορφία. Μ' αρέσουν οι δανειστικέ ταινίε. Μ' αρέσουν πολύ οι ταινίε στο σινεμά, οι ιδανικές. Τα, τις έχω δει αυτές τις ταινίες το εθνικό κανάλι της Εστονίας και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Ξέρω ότι έχετε πολύ καλές ταινίες στην ε, Δανία. Αυτοί όμως οι οποίοι είναι οι διανομής ταινιών δεν έχουν πάρει πολλές ταινίες από τη Δανία. Τι θα κάνει ένας άνθρωπος σαν και εμένα λοιπόν πρέπει να έχουμε διαμεθοριακή πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο. Είμαι έτοιμο να πληρώσω γιατί θα ήθελα να δω αυτέ τι ε, δανεικές ταινίε. Αυτό θα πει πολιτιστική πολυμορφία. Όταν υπάρχει πρόσβαση λοιπόν σε αυτά τα αριστουργήματα. Αυτό θα πει πολιτιστική πολυμορφία. Πρόσφατα είχα συναντήσει ε, το διευθυντή ενός μιας γερμανικής ταινιοθήκης. Μου είπε ότι είναι εκατοντάδες πολύ καλών ταινιών σε ψηφιακή μορφή ήδη, αλλά οι διανομής ταινιών δεν ενδιαφέρονται να πάρουν άδειε για αυτές τις ταινίες επί τη βάση της εδαφικότητας για να προβάλλουν αυτές τις ταινίε εδώ στο Βέλγιο. Γιατί δεν έχουν οικονομικό κίνητρο να το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω τώρα σε όλο τον κόσμο. 100.000, ένα, ένα εκατομμύριο, δέκα εκατομμύρια ανθρώπων που θέλουν να δουν αυτές τις ταινίες, αλλά δεν βρίσκονται όλοι στην ίδια χώρα. Ποια είναι η λύση λοιπόν για να έχουμε διαμεθοριακή πρόσβαση. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Θα πρέπει να μπορούμε να πάρουμε τα χρήματά τους και η πρότασή μου είναι ακριβώς να εξασφαλίσουμε τη διαμεθοριακή πρόσβαση. Με αυτή την πρόταση εγώ υποστηρίζω και την δημιουργία καλύτερου πολιτιστικού περιεχομένου, καλύτερων ταινιών, μεγαλύτερης πολιτιστικής ε, πολυμορφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παγκόσμιοι λοιπόν παίκτες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και τις 28 αγορές της Ευρώπης. Αλλά η εθνική παραγωγή είναι στα δύσκολα. Δεν μπορούν να πουλήσουν την παραγωγή τους, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις διαφορετικές ρυθμίσεις σε 28 χώρες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματική φραγμή, αυτή είναι η πραγματική δυσκολία για να προστατεύσουμε την πολιτιστική πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, ετέθηκε το ερώτημα για τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Αλλά δεν είμαι έτοιμο εδώ να προτείνω συγκεκριμένα εργαλεία. Εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως να επισημάνουμε τους κύριους τομείς όπου υπάρχουν προβλήματα και θα εργαστούμε για τους τομείς αυτούς και θα ήθελα να προτείνω μια σειρά από νομοθετικές πράξεις και μη νομοθετικές πράξεις σε επίπεδο κανονισμών σε ρυθμιστικό πλαίσιο μάλλον ώστε μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και μετά θα συζητήσουμε τι είδους εργαλεία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και όλες αυτές οι λύσεις θα βασίζονται σε αξιολόγηση αντικτύπου και στα αποτελέσματα των δημοσίων διαβουλεύσεων και τα λοιπά. Είναι πολύ νωρίς λοιπόν να σας πω σήμερα τι είδους συγκεκριμένα εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε. Αν θα προτείνουμε μια νέα οδηγία ή κάτι διαφορετικό. Λυπάμαι. Αυτά. Δεν τα έχω αυτά τα εργαλεία ακόμα. και τα πακέτα. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι όπως τα λένε οι επιχειρηματίες είναι βασικός φραγμός η υψηλή τιμή όσον αφορά την ε, αποστολή των πακέτων. Είναι φραγμός για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ένωση. Όλοι ξέρουμε ότι οι τιμές αποστολής των δεμάτων πρέπει να εξαρτάται από το κόστος. Όμως, στην πραγματικότητα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζουν. Όλοι ξέρουμε ότι όσο με το πρίστον οι τιμές διαμορφώνονται από το τελευταίο μίλι γιατί εκεί είναι η πιο μεγάλη δαπάνη. Στην πραγματικότητα όμως, να, ας την Πολωνία για παράδειγμα. Μία αποστολή από Βέλγιο προς Πολωνία. Μιλάω για δέμα 2 κιλών. Θα πάει στα 26 ευρώ. Όμως από την Πολωνία προς το Βέλγιο 14, κάτι, 14, 30, ακόμα 40. Όμως φυσικά οι μισθοί, τα εργατικά είναι πολύ πιο φθηνά στην Πολωνία παρά στο Βέλγιο. Όμως το, το κόστος από τη χώρα που κοστίζει ε, τα εργατικά κοστίζουν λιγότερο προς την πιο ε, ακριβή χώρα είναι κάτι που κοστίζει πολύ λιγότερο για τα θέματα παρά το αντίστροφο. Και επομένω το ερώτημα είναι γιατί. Α, για τη Δανία. Να πάρουμε πάλι παράδειγμα. Τη Δανία και τη Σουηδία. Πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει κανεί γιατί. Η αποστολή από την μία χώρα στην άλλη κοστίζει 27 ευρώ και από μια άλλη προς την πρώτη χώρα τα, ίδια δύο κιλά πάνε στα 42 ευρώ και μιλώ μάλμα στην Κοπενχάγη δηλαδή για κάποιες πόλεις που είναι πάρα πολύ κοντά μία στην άλλη όπου η απόσταση δεν είναι καθόλου μεγάλη οπότε και εγώ ίδιος Όταν μετακόμισα, παράγγειλε ένα χαλί, δύο επί τρία. Το παράγγειλε από τη Γερμανία. Και πλήρωσε για να μου το φέρουν σε πακέτο 80 ευρώ. Ένα χαλάκι, δύο επί τρία. Μα, ε, κοιτάξτε, θέλουμε τα για δύο κιλά από το μάλλον στην Κοπεχάγη. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Δεν θέλω να αρχίσουμε να νομοθετούμε για την τιμολογική πολιτική, αλλά θέλουμε να γνωρίζουμε από πού προέρχονται, από πού διαμορφώνονται αυτές οι τιμές. Έχουμε και αυτή την οδηγία για τις καθολικές υπηρεσίες. Είσαστε έτοιμοι να ξανανοίξουμε τον ασκό του αιώλου για αυτό το πράγμα, για αυτή την οδηγία. Ε, μήπως όμως πρέπει να το κάνουμε, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, οι εξελίξεις είναι εντυπωσιακές, 15 20% την ημέρα σε πρώτες τιμές για αυτές. Όμως, μόλις την η εβδομάδα, είχαμε μια συνάντηση με το κρατικό τοχυδρομείο και τα βλέπανε αισιόδοξα τα πράγματα και λέγανε ότι τα δέματα εκείνα αντισταθμίζουν την μείωση του κόστους των τελών τέλο πάντων αποστολής γράμματος. Είδε λοιπόν καλά τα έχουν πάει μέχρι τώρα τα δέματα. Όμως Υπάρχουν παράπονα για την έλλειψη της διαφάνειας. Και σε σχέση με την ανίγνευση παρακολούθηση της πορείας του δέματος εδώ στα περισσότερα κατημέλη ήδη τώρα έχουμε αυτή την υπηρεσία, αυτό το σύστημα παρακολούθησης. Σύστημα το οποίο μας δίνει να καταλάβουμε που βρίσκονται τα δέματα. Και αν τυχόν βρίσκονται εκεί που δεν έπρεπε. Ευτυχώ, ευτυχώ που, το, που έχουμε αυτή την υπηρεσία. Δεν κατηγορώ τα ταχυδρομεία. Θέλω να σα πω ότι παρά τι δυσκολίε, καλά τα πάνε. Να κάτι ρώτησε ο Γιος Κάλλας. Άλλο. Για τον κανονισμό καλύτερη λύση είναι να μην υπάρχει καθόλου κανονισμός. Αν δεν υπάρχει λόγος, δεν χρειάζεται να νομοθετήσουμε. Βέβαια, καμιά φορά υπάρχουν κάποια γενικά προβλήματα τα οποία μας αγκαλούν να παρέμβουμε. Επίσης θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και όσον αφορά τις καινοτομίες μέσω του διαδικτύου. προσοχή γιατί όταν ε, νομοθετούμε πολλές φορές σκοτώνουμε την γενοτομία, άρα θέλει μεγάλη προσοχή. Να νομοθετούμε μόνο όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη προς τούτο. Ξέρετε όλοι τι πιστεύω για το Ρώμη. Για τη χρέωση του Ρώμη. Της περιαγωγής. Όλοι θα πρέπει τις υποσχέσεις να τις στήρουν. Και, κατά την προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογέ, όλα τα κόμματα υποσχέθηκαν μείωση αυτών των τελών. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα να τηρηθούν τα υπεσχημένα. Άρα μια σωστή πρόταση θα ήταν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, να ξεκινήσουν τρι, τριμερείς διάλογοι με, με κοινοβούλιο ε, και μας και τα κρατημέλη. Να καταργηθούν τα επιπρόσθετα τέλη για την ε, περιαγωγή. Όμως τα πράγματα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι το ικανοποιητικό αυτό το 5 συν 5 συν 5. Γιατί στους ψηφοφόρους υποσχεθήκαμε κατάργηση των προσθέτων τελών. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μα και την εκτίμησή μα προ τον Επίτροπο για τον χρόνο του σήμερα το απόγευμα. So, and I, I'm, ready to be here. Μάλιστα. Και πάλι είμαστε εδώ, λοιπόν. Θα ξανάρθω όποτε με θέλετε. Θα σας καλέσουμε σύντομα, επιτροπέ. Όχι την άλλη Παρασκευή, πάντως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Και τώρα περνάμε στο επόμενο τμήμα τη σημερινή σας διάταξη για τον προπολογισμό. Και βλέπω ότι είναι εδώ η ηγητή μα. Εξαιρετικά. Υπάρχει υπάρξει ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα λοιπόν... Έχουμε και τον κύριο Φερνάντες εδώ, εξαιρετικά. Και την κυρία Γκάλε από την ΕΜΚΟ και τον κύριο Φερνάντες. Ποιο θα ήθελε να πάρει το πρώτο στο λόγο, ο κύριο Φερνάντες. Πολύ ωραίο, ναι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι συντομότατο. Ναι. Οι κατευθυντήρες γραμμές του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ήδη εγκριθεί. Εγκρίθηκαν λοιπόν από την Ολομέλεια. Δεν είμαι εμπειρογνώμων τώρα για τα θέματα της Επιτροπής σας. Απλώς έρχομαι για να ακούσω τις απόψεις σας, τις προτεραιότητές σας, τα θέματα τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 2016. Ε, εμείς έχουμε τις προτεραιότητες σε τρία ε, στα αγγλικά βέβαια. Απασχόληση, επιχειρήσεις και το επιχειρήν, το πνεύμα του επιχειρήν. Για να γίνει αυτό όμως γεγονός, χρειαζόμαστε μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση των προγραμμάτων τα οποία μπορούν να συμβάνουν προς την επίτευξη αυτού του, στο, του στόχου, προγράμματα όπως το COSME, το έρασμο συν, ο ορίζον 2020, η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Αυτά πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Για μας είναι απαραίτητη η αλληλεγγύη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα ταμεία συνοχής, η εξωτερική αλληλεγγύη. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα γύρω από την Ευρώπη και το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη. Η εξωτερική αλληλεγγύη είναι η κατηγορία 4 που έχουμε στην ανθρωπιστική βοήθεια και έχουμε επίσης και τα θέματα ασφαλείας που συνδέονται με αυτές τις δύο προτεραιότητες. Ξεκινάμε από την αρχή ότι τα προβλήματα για τις πιστώσεις πληρωμών θα λυθούν το 2015 και το Συμβούλιο συγκεκριμένα θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις του και τις δεσμεύσεις του. Στα πλαίσια λοιπόν της Επιτροπής σας θα ήθελα να μιλήσω για το χρονοδιάγραμμα. 25 Μαΐου προβλέπεται η Κομισιόν να παρουσιάσει το προσχέδιο προϋπολογισμού, κάτι το οποίο είναι σημαντικό, ιδίως γιατί η Επιτροπή είναι το εξή. Είναι οι προπαρασκευαστικές δράσεις και τα πιλωτικά σχέδια. 4 Ιουνίου είναι η καταληκτική προθεσμία για να παρουσιαστούν νέα πιλωτικά σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις. 17 Ιουνίου θα πρέπει να εγκριθούν οι εκθέσεις, σχετικά 3 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για τον προϋπολογισμό και στα μέσα Σεπτεμβρίου θα γίνει η έκθεση των ψηφισμάτων για τον προπολογισμό. 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. 12, 13 Οκτωβρίου ψη... ψηφοφορία στην Ολομέλεια και μετά η διαδικασία συνδιαλλαγής μεταξύ 29 Οκτωβρίου και 18 Νοεμβρίου. Επιμένω για το θέμα των πιλωτικών σχεδίων αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη τέτοια, τέτοια, τρία τέτοια σχέδια, δύο πιλωτικά και μία προπαρασκευαστική δράση. Έχουμε ένα νέο πιλωτικό σχέδιο, το οποίο ξεκίνησε φέτος. Για την Επιτροπή σας έχουμε το πρόγραμμα δράσης για τα τελωνία, που εφέτος είδε μία αύξηση κονδυλίων σε σχέση με το 2014 και για την ε, σχεδίαση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου προτείνεται και πάλι το 2016 μια αύξηση αλλά το σχέδιο προϋπολογισμού της Κομισιόν δεν θα παρουσιαστεί παρά μόνο 27 Μαΐου. Για τα προγράμματα που αφορούν τον καταναλωτή, κατηγορία 3, το πρόγραμμα αυτό υπέρ των καταναλωτών έτυχε αύξηση στο 2015 σε σχέση με το 2014. 0,6 εκατομμυρίων ευρώ και για το 2016 προβλέπεται μία αύξηση σε ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τις στόχους αυτούς. Όπως όμως καταλαβαίνετε, θα δω να σας δώσω αυτές τις πληροφορίες, αλλά και για να ακούσω ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες, γνωρίζοντας ότι αν βάλουμε στον προϋπολογισμό όλα αυτά που θέλουν οι επιτροπές, θα χρειαζόμασταν ένα προϋπολογισμό πολύ πιο διωγγωμένο από αυτά που είναι τα όρια μας και ξέρετε τα όρια μας είναι περίπου το 1% του, ε, του ΑΕΠ ή ΑΕΧ της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν ήταν αυτά που ήθελα να σας αναφέρω και φυσικά θέλω να συνεργαστώ μαζί σας για να πετύχουμε τον καλύτερο δυνατό προϋπολογισμό που να λαμβάνει υπόψη και τις δικές σας προτεραιότητες. Σας ευχαριστώ και με άλλη χαρά και βοήθεια που είσαστε εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πλητικό μας πρόγραμμα πέρσι εστιάστηκε στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δώσω το λόγο τώρα στο δικό μα εισηγητή. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. σα ευχαριστώ, κύριε Φερνάνδες. Θα μιλήσω γκουικά. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φερνάνδες για το γεγονό ότι ήρθε εδώ στην Επιτροπή μα και μας πληροφόρησε για τα πιο σημαντικά στοιχεία, τα οποία τα γνωρίζουμε ουσιαστικά γιατί, όπως είπατε και στην προηγούμενη ολομέλεια, ψηφίσαμε. Και έτσι ε, ρυθμίστηκαν κάποια θέματα δομής. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια καταρχάς για τη δομή αυτή ακριβώς. Ως ε, μέλος της Επιτροπής ΙΜΚΟ, Πρέπει να πω ότι μου λείπει κάτι από την δομή αυτή και αυτό που λείπει είναι η εσωτερική αγορά. Βλέπω λοιπόν ότι κοιτάμε θέματα πιο πολύ, σε, πιο πολύ επενδύσεων. Αυτή είναι η βασική κατεύθυνση, το βασικό ζήτημα, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω και το εξή. Να μην ξεχνάμε κάποια συγκεκριμένα θέματα τα οποία φροντίζουν και εγγυώνται την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρατε. Μιλήσατε για την ε, ενιαία αγορά, την προστασία του καταναλωτή για την ε, πλήρη ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Πόσο μάλλον επειδή η ίδια η ενιαία αγορά έχει από μόνη της ε, πολιτική αξία. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν ε, πολιτικό τομέα για όλους μας και θα πρέπει να παραμείνει έτσι. Είναι σημαντικό λοιπόν για την ε, ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία ενιαία εσωτερική αγορά και αυτή η εσωτερική αγορά θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Και περνάω λοιπόν στο βασικό ζήτημα στις προτεραιότητές μας. Μία από τις πιο βασικές μας προτεραιότητες είναι η πολιτική του καταναλωτή. Πρόκειται για μία προτεραιότητα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι έχουμε επαρκή μέσα για τους σκοπούς αυτούς και ότι θα πρέπει να διαθέσουμε τα μέτρα αυτά, τα μέσα αυτά. Καλά λάβει χώρα λοιπόν σχετική το σχετικό εγχείρημα. Χρειαζόμαστε έναν προπολογισμό ο οποίος θα διασφαλίσει ότι η προστασία του καταναλωτή ότι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή θα αυξηθεί και ότι μπορούμε να είμαστε πραγματικά έμπιστοι γιατί προστατεύουμε τα συμφέροντα του καταναλωτή. Ε, θα πρέπει επίσης να διατεθούν ε, μέσα για την ευθύη ανάπτυξη και για σκοπούς απασχόλησης, θέσεων απασχόλησης. Άλλη μία προτεραιότητα είναι η Τελωνιακή Ένωση, η καταπολέμηση της απάτης επίσης. Στον τομέα αυτό, για να είμαστε αποτελεσματικοί, χρειαζόμαστε ίσως ε, περισσότερα μέσα. Και γιατί αναφέρω συγκεκριμένα την καταπολέμηση της απάτης. Δεν είμαι βέβαιη ότι εκεί που αναφέρατε την Τελεωνιακή Ένωση, συμπεριλαμβάνεται και την ε, καταπολέμηση της απάτης. Πιστεύω ότι στην παρούσα φάση θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε και το Single Market Forum. Μία άλλη προτεραιότητά να αναφέρω, μία πλατφόρμα για την ε, εναλλακτική επίλυση διαφορών. Πρόκειται για ένα εργαλείο για την αποτελεσματική επίλυση διαφορών. Αυτό στην ενιαία αγορά λοιπόν θα μπορούσε να επιλύσει σημαντικές διαφορές που ενδεχομένως να οδηγούσαν σοβαρά προβλήματα. Έχω κάνει λοιπόν ένα σχέδιο το οποίο και θα εξετάσουμε στην Ειδική Επιτροπή, στην Αρμόδια Επιτροπή στις αρχές Μαΐου και εννοείται πιο λεπτομερή ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Ε, τον εισηγητή μας θα ήθελα τώρα να ρωτήσω αν υπάρχουν συντονιστές ή σκιώδες εισηγητές οι οποίοι θα θέλουν να πούνε κάτι. Η Ντάνα, ο Ντάν μάλλον πρώτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Η βασική μας αρχή στον προϋπολογισμό είναι πάντα η ίδια. Σε γενικές γραμμές εμείς δεν θα υποστηρίξουμε ποτέ αυξήσεις ε, σε δαπάνες ή νέα πιλωτικά σχέδια εκτός αν υπάρχει κάποια τεκμηριωμένη ανάγκη για όλα αυτά και εκτός αν μπορούμε να βρούμε άλλες περικοπές σε άλλα τμήματα του προϋπολογισμού. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιούνται τα λεφτά των φορολογουμένων χωρί αποχρόντα λόγο. Αλλά θα εξετάσουμε τα πιλωτικά προγράμματα και αν υπάρχει πραγματική ανάγκη μπορούμε να τα υποστηρίξουμε. Αλλά γενικά θέλουμε να πετύχουμε και περικοπές σε άλλα, αντίστοιχε περικοπέ σε άλλα σημεία του προπολογισμού μα το προπολογισμό δεν χρησιμοποιείται χρησιμοποιείτε τα ποσά, τα χάνετε. Επομένω. τα χρήματα αυτά, ό,τι δεν χρησιμοποιήσουμε για την έννοια αγορά, θα τα χάσουμε. Μόνο πέρυσι το κατάλαβα αυτό. Είναι ένα ποσό για τις, ε, την εσωτερική αγορά που δεν μπορεί να πάει αλλού. Ναι, θέλω να επανέλθω, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αν όλες οι επιτροπές κάνουν το ίδιο και δεν χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά, κάνουμε μια εξοικονόμηση. Μα θα φύγουν τα λεφτά και κάποια πράγματα δεν θα μπορείτε να τα κάνετε. Ξέρω ότι εσείς δεν θέλετε πιλωτικά προγράμματα, αυτό είναι δικαίωμά σας, αλλά στην Επιτροπή μας αυτή παίρνουμε πολύ σοβαρά την ευθύνη μας να υποστηρίξουμε πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, χωρίς μικρόφωνο μιλητής. Κάποιος θέλει να λάβει το λόγο, κύριο Κουέλιου. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Φερνάντζης και την πρότασή του. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω αυτό το οποίο μας είπε ήδη ο εισηγητής μας. Είναι πολύ καλό για μας στην Επιτροπή μας να καταλάβουμε ότι ο εισηγητής υποστηρίζει την ανάγκη της υποστήριξης του επιχειρήν, των, της επιχειρήσης και την απασχόληση. Δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν ο εισηγητής του Γενικού Προϋπολογισμού να έχει ευθυγραμμιστεί με τις δικές μας προτεραιότητες. Αυτό θέλω να το αναγνωρίσω. Και επίση: να τονίσω τον ρόλο των προπαρασκευαστικών δράσεων και των πιλωτικών σχεδίων. το, τα κονδύλια για την εκπαίδευση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων για τον ψηφιακό κόσμο είναι μια περίπτωση που μπορούμε εκεί πέρα να βελτιώσουμε τα πράγματα, να κάνουμε τη διαφορά. Δεν μιλάμε για μεγάλα χρηματικά ποσά. Μιλάμε για τη δυνατότητα να υπάρχει καλύτερη χρήση κονδυλίων μικρού όγκου που μπορούν να βελτιώσουν πολύ τα πράγματα. Όπως είπε και ο κύριος Φενάντες, έχουμε καιρό μέχρι 4 Ιουνίου για να κάνουμε προτάσεις για το 2016 στον τομέα αυτό. Αλλά θα ήθελα από τώρα να πω ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε να κάνουμε προτάσεις στον τομέα των καταναλωτών. Στην ε, προστασία των καταναλωτών όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα να τα υποστηρίξουμε. Ευχαριστούμε για όσα μας είπατε, λέει η κυρία Στάιλερ. Άλλοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Κοιτάω γύρω γύρω. Μήπως θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο. Όχι. Καλώς. Μου είπα να σας ρωτήσω. Μπάς και θέλατε. Καλά. Θέλει να δευτερολογήσει ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστούμε. Oui, je Ναι, να σας ευχαριστήσω για τα όσα είπατε. Συνάδελφοι, και θα ήθελα να τονίσω ότι έχει ήδη καταβάλει μεγάλη προσπάθεια και έχει προχωρήσει στη δουλειά που θέλουμε να γίνει η συγκίτρια. Και επίσης δεν θέλω να ξεχνούμε ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης όχι, όχι δεν λέμε το κοινοβουλίο που είναι μικρότερος, αλλά της Ένωσης ο προϋπολογισμός είναι περίπου 1%, 1 του ΑΕΧ. Το ΑΕΠ μάλλον, 20% είναι στη ΣΥΠΑ το αντίστοιχο ποσό. Και μιλούμε για 94% του προπολογισμού το οποίο πηγαίνει σε επενδύσεις. Μόνο 6% αφορούν τις δαπάνες λειτουργίας, ε, τις διοικητικές δαπάνες. Να, ένα προπολογισμό που δίνει προσθεμένη αξία. Και για κάποια κρατή μέλη μιλούμε για το 50% των κρατικών αναπενδύσεων. Και βεβαίω. πρέπει να πιάνουν τόπο αυτά τα χρήματα. Επίσης, θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι παρά το ότι τρέχουμε 28 κράτη-μέλη και νέα κατανομή αρμοδιοτήτων παραμένει ο προϋπολογισμός 1% του ΑΕΠ. Τόσο να αφορά αυτή την εύστοχη ερώτηση για την ιστορική αγορά. Μπορεί να βοηθήσει ο προπολογισμό. Νομίζω έχετε αναλάβει και την έκθεση για το σχέδιο Γιούγκερ. Να, πώς ενισχύεται και υποστηρίζεται η ιστορική αγορά τώρα για τις επενδύσεις, για, το ψηφιακό θεματολόγιο, εναρμόνιση και υποστήριξη. Πολύ σημαντικά. Συμφωνώ τις που είπατε, για τους καταναλωτές δηλαδή, και εδώ ωφελεί η ιστορική αγορά και να μην ξεχνούμε ότι είμαστε 500 εκατομμύρια εν δυνάμει καταναλωτών εδώ. Αν θυμηθείτε την Τελωνική Ένωση που είχαμε 15% των ε, δασμών και λοιπά του Κοινοβουλίου. Πολύ σημαντικά αυτό το ποσά για τον προπολογισμό. Επίσης έχουμε και την καταπολέμηση της απάτης. Και αυτή είναι μια προτεραιότητα. Τώρα η δυνατότητα να υπάρξουν πλατφόρμες για την επίλυση των διαφορών, να δούμε αν αυτό γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος για τους καταναλωτάς. Όμως, ακόμα δεν μπορώ τίποτα. Δεν μπορώ να σας πω. Τι πρεκοδοτήσεις θα προβλέπονται. Είπαμε εκεί στη δράση για τα τελωνία ότι κάτι προβλέπεται στα πλαίσια του, του, του, του πλαισίου. Έχουμε 71,8. Και επίσης έχουμε και στο τρίτο κεφάλαιο το πρόγραμμα τους καταναλωτές και εκεί προβλέπονται 25,9 εκατομμύρια. Οπότε να δούμε τι θα προτείνει η Επιτροπή. Και επίσης να δούμε πώς θα τρέξουν αυτά τα πιλωτικά προγράμματα που έχουν σχέση με την προπαρασκευαστική δράση που ήδη έχει αρχίσει να εξελίσσεται, να λειτουργεί. Ευχαριστώ για την βοήθειά σας, αλλά και για την ενημέρωση και για τις προτεραιότητες. Να ξέρετε ότι θα δώσω τη μάχη μου με την έκθεση. Και ε, κάπου θα τα πούμε, κάπου θα συνδεθούμε. Ε, και αν δεν τα πούμε από κοντά, τότε θα μάθω τις προτάσεις σας, από τις ε, τροπολογίες τις οποίες θα έχετε υποβάλει και εγκρίνει. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Φερνάντες που ήρθατε 24 Απριλίου για μετάφραση, συζήτηση 6 και 7 Πέμπτου για τροπολογίες 12 Μαΐου, ψηφοφορία εδώ 4 Εκτού και έγκριση και για τα πιλωτικά μαζί και για τους προπολογισμούς 17 Ιουνίου υποβολή εκεί. Πάμε τώρα τα στο τελευταίο θέμα της μέσης διάταξης. Είναι η έκθεση για τα προϊόντα από φώκες. Κριστιαν Μπουσόη λέγεται ο εισηγητής μας, ο οποίος έχει τη σκητάλη. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Στάιλερ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, τους σκιώδεις εισηγητές και το προσωπικό της ε, γραμματείας Τη Επιτροπή ΣΥΜΚΟ για τη βοήθειά του την τελευταία εβδομάδα και τι προσπάθειε που έχουν καταβάλει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο πάρα πολύ χρονικά σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Προσβλέπουμε στο να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση μέχρι τον ε, Ιούνιο και θέλω να ευχαριστήσω το, τους συντονιστές και το, την Πρόεδρο για το γεγονός ότι δέχτηκαν αυτό το χρονοδιάγραμμα. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι μετά από τι συναντήσεις που είχα με εκπροσώπους του Δανικού και Γρυλανδικού Κοινοβουλίου, με ΜΚΟ και την Κομισιόν, πιστεύω ότι το κυνήγι που κάνει των φωκών, των Ινουίτ και άλλων ε, ηθαγενών κοινοτήτων δεν θίγει το οικοσύστημα που, όπου ζουν οι φώκες και ούτε οδηγεί σε βάρος για το περιβάλλον. με τον οποίο μπορούν να διατηρήσουν τις κοινότητές τους και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους. Χρειάζονται τροφή από τις φώκες, αυτό είναι τμήμα της πελτιστικής τους παράδοσης και έχουν κάθε σεβασμό για την ευζοία των ζώων. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ε, κυνηγούν φώκες για λόγο οικονομικής εκμετάλλευσης και δεν κυνηγούν ε, ανήλικα ζώα. Η πρόταση αυτή λοιπόν, όπως ξέρετε, έχει, έχει κάποιο πολιτικό βάρος, αλλά ο στόχος της είναι να εφαρμόσει τις συστάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου από τον προηγούμενο Ιούλιο σε σχέση με τον βασικό προκανονισμό 2009 το εμπόριο σε προϊόντα που προέρχονται από φώκες. Είναι και η νομική, δίνει και μία νομική βάση για να μπορέσει ο αρμόδιος κανονισμός του 2010 να τεθεί σε συμφωνία με τις αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η Κομισιόν λοιπόν έχει υποβάλει αυτή την πρόταση για να συμμορφωθεί η νομοθεσία με την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν την Κομισιόν για την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει και την καλή συνεργασία και τον καλό διάλογο. Θέλω να τονίσω επίση ότι και η πρότασή μα προήλθε από την πρόταση τη Κομισιόν με μία μικρή καθυστέρηση. Δεν υπάρχει εδώ κάποια έκθεση αντικτύπου για την νομοθεσία αυτή, ούτε κάποια έκθεση για εφαρμογή όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 της νομοθεσίας. Αν λάβουμε υπόψη λοιπόν ότι ο νέος κανονισμός έχει στόχο να εφαρμόσει την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σε σχέση με τον κανονισμό του 2009 για το εμπόριο σε προϊόντα που προέρχονται από φώκες, σύμφωνο με την ε, ε κατάρριξη της εξαίρεσης MRM. Θα ήθελα όμως εδώ να έχω την άποψη των εισηγητών και της Κομισιόν αν υπάρχει δυνατότητα να προβληθεί και πάλι μια νέα εξαίρεση και αν αυτή θα έρθει σε σύγκρουση με την απόφαση του ΠΟΕ. Σε ό,τι αφορά την εξαίρεση IC, έχω λάβει υπόψη την πρόταση της Κομισιόν, λαμβάνοντας υπόψη και το δικαίωμα της ε, αυτοδιάθεσης των Ινουίτ και άλλων ηθαγενών κοινοτήτων. Επομένως, η πρότασή μου επαναλαμβάνει ότι η θύρα φωκών είναι βασικό στοιχείο της κουλτούρας και της ταυτότητάς τους και είναι απαραίτητη για την επιβίωσή τους, τους δίνει τροφή και εισόδημα για να μπορέσουν να διατηρηθούν οι ηθαγενείς κοινότητες διατηρώντας τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους και διατηρώντας την πολιτιστική τους κληρονομιά. Με τη βοήθεια της νομικής υπηρεσίας προσπάθησε να ξεπεράσω τη σύγκρουση μεταξύ του άρθρου 3.5 και του άρθρου 3.1 που υπήρχε στο αρχικό κείμενο της πρότασης της Κομισιόν. Πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει κατεξουσιοδότηση πράξη για να περιορίσει τον όγκο των προϊόντων φώκια στην αγορά μόνο όταν τα στοιχεία μας δείχνουν ότι ο αριθμός των φωκών που έχει κυνηγηθεί έχει θηρευτεί η ποσότητα των πλεοριόντων μπορούν να καταδείξουν ότι το κυνήγι γίνεται για εμπορικούς και μόνο Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επάγρυπνοι και να γνωρίσουμε ότι είναι πολύ δύσκολο και ιδιαίτερα δύσκολο να καταλάβουμε πότε μια παραδοσιακή κοινότητα περνάει από απλώς ε, επιβίωση σε εμπορικές θηρευτικές δραστηριότητες. ό,τι αφορά το σημείο 6 για την άδεια θύρας, θεωρώ ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολλές δυσκολίες για την καναδική πλευρά και μπορεί να ερμηνευτεί και ως διάκριση με την συμφωνία λοιπόν των συναδέλφων μου, των σκιωδών συγητών, θεωρώ ότι πρέπει να επαναδιατυπωθεί τονίζοντας ότι η θύρα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την ευζοία των ζώων. Το νέο άρθρο το οποίο έχει προταθεί το 5α σε σχέση με την ανάγκη να είναι σωστή η πληροφόρηση όλων των πολιτών σε σχέση με τα προϊόντα από φώκες που έρχονται από την κοινότητα των Ινουίτ και άλλες ηθαγενείς κοινότητες έχουν νομικό χαρακτήρα και είναι πολύ σημαντικά. Το να υπάρχουν εκστατείες για μεγαλύτερη συνειδητοποίηση που θα πληροφορήσουν τον πληθυσμό για τα θέματα αυτά μπορούν να γίνουν και επί τη βάση του στόχου 2 του κανονισμού για την πληροφόρηση των καταναλωτών. Αλλά αυτό δεν πρέπει να αφορά τα προϊόντα από φώτιες, αλλά για να γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι είναι ηθικά προϊόντα, είναι δεοντολογικά παραχθέντα προϊόντα. Κλείνω την παρέμβασή μου λέγοντα ότι ο λόγος για την τροποποίηση του άρθρου 7 είναι ότι είδαμε ότι η διαδικασία αναφορών δεν ήταν αρκετά αντικειμενική και δεν σεβόταν τα κριτήρια του άρθρου 7 του κανονισμού. Πιστεύω ότι για τον τελικό κανονισμό η Κομισιόν θα πρέπει να αξιολογήσει τον αντίκτυπο για το κοινωνικό ε, συμφέρον των Ινουίτ και άλλων κοινοτήτων μεταξύ των οποίων και το δικαίωμά τους να έχουν τρόφιμα και εισόδημα για να μπορέσουν να διατηρήσουν την ζωή τη κοινότητά του. Και τέλος. Να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή και τους άλλους συναδέλφους ε, που μοιράστηκαν τις απόψεις τους μαζί μου και που ε, ενδιαφέρθηκαν να ακούσουν και τι είναι δικέ μα απόψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει κύριε Πρόεδρο. Και τώρα να ακούσουμε του κοιόδε. Η κυρία Σοντεμόζα από του Σοσιαλιστέ Δημοκράτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω δανέζικα και το είπα και προηγουμένως, αλλά αυτή θα μιλήσω όλα δανέζικα. Να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Σε ό,τι αφορά την απαγόρευση της εξαγωγής ε, των προϊόντων αυτών, ε, είναι κάτι που μας απασχολεί εδώ και καιρό και ήμουν ήδη το 2008 εισηγήτρια από την ομάδα μας και όπως και τότε πιστεύουμε ότι είναι καλό να παραμείνει η απαγόρευση για τις φώκες αυτές, για τα προϊόντα φώκες, για τα πολύ νεαρά ζώα και σε ό,τι αφορά και τον τρόπο θύρευσης. Αυτή είναι η θέση των συλλεκτών και Δημοκρατών. Αυτό δεν είναι όμω το θέμα τη σημερινή συζήτηση, όπω ανέφερε και ο εισηγητή. Θέλουμε να δούμε πώς η απόφαση αυτή του ΠΟΕ μπορεί να εφαρμοστεί. Και υπήρχε και αυτή η εξαίρεση για τους Ινουίτε. Είναι σημαντικό λοιπόν να πούμε δύο λόγια για το θέμα αυτό, γιατί όπως είπε ο εισηγητής, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτή οι τρόποι αλίευσης, θύρευσης, ε, δεν προκαλούν πρόβλημα σε ό,τι αφορά την κοινότητα των ασκημών. Ο τρόπος που αντιδρούμεται στην ε, απόφαση αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι οι Ινουίτες και οι άλλες φυλές θα πρέπει να έχουν μια δυνατότητα ε, χρήσης και θύρευσης των προϊόντων αυτών για να επιβιώσουν. Αυτό συνάδει άλλωστε και με τα καλά πρότυπα σε ό,τι αφορά τα ζωά με σχετική συμφωνία της Greenpeace, η οποία συμφωνεί με τον τρόπο αυτό θύρευσης από πλευρά των Μενουιδών. Θεωρεί ότι συνάδει με τα φυσικά πρότυπα και με τα πρότυπα τα οποία ισχύουν. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι σημαντικό εδώ στο Κοινοβούλιο να δώσουμε την δυνατότητα να συνεχιστεί η εξαίρεση αυτή ως εξαίρεση πραγματικά να λειτουργήσει ως εξαίρεση, να συνεχίσει να υπάρχει δυνατότητα να συνεχιστεί η θέρευση φώκιας ε, για λόγους επιβίωσης. Το μεγαλύτερο τμήμα των ε, τροπολογιών που έχει υποβάλει ο εισηγητής μας βρίσκουν σύμφωνος. Σε κάποιε περιπτώσει πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να βρούμε μια διαφορετική διατύπωση σε ό,τι αφορά το σημείο 6, την τροπολογία 6, μιλάτε για προκλήσει. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια μικρή αναδιατύπωση. Το βασικό είναι να μην περιοριστεί η εξαίρεση αυτή, αλλά να συνεχίσει να ισχύει. Ε, ως εκ τούτου ενδεχομένω να καταθέσω και εγώ τροπολογίες για το, τη διευκρίνηση του ορισμού της ε, θύρευσης φώκιας. Εδώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει κάποια βελτίωση ελαφριά σε σχέση με αυτά που προτείνει ο εισηγητής. Αντιμετωπίζουμε και προβλήματα Θα είχαμε προβλήματα στην Ευρώπη αν καταργούσαμε το κυνηγήφό φώκια εντελώ. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν μια νέα διατύπωση για το ότι σεβόμαστε τις, ε, τα πρότυπα που έχουν ε, καθοριστεί ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όμως και στη βαλτική τα αλλιευτικά αποθέματα θα πρέπει να συνεχίσει να επιτρέπεται η αλλιεύση και θα πρέπει όλα αυτά φυσικά να γίνουν μετά από προσεκτική εξέταση. Ε, Επίση, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι υποστηρίζω κατά 100% την διεξαγωγή μελέτη αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιε είναι οι συνέπειε τη νομική ρύθμιση αυτή. Υποστηρίζω λοιπόν επίση 100% την ενημερωτική εκστρατεία, προκειμένου οι Ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίζουν ότι τα προϊόντα φώκια ε, παράγονται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές ε, διατάξεις και ανταποκρίνονται στα σχετικά πρότυπα. Θα συνεχίσουμε τη συνέχεια συνεργασία με τον εισήγητη και με βέβαιη ότι θα προκύψει ένα ε, εγγραφό καλό σε ποιότητα μέσα στα χρονικά πλαίσια. Ευχαριστώ του Ισιάτορα, ο κ. Τάντον. Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή γιατί ανέλαβε το θέμα αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα και δεν έχουμε πολύ χρόνο για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Νομίζω ότι οι προτάσεις σας είναι πολύ καλές και λαμβάνουν υπόψη πολλά από τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε από τη δική μας άποψη. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να συμμορφωθούμε προς τις αποφάσεις του ΠΟΕ. Αυτό είναι γενικό σε συνολικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τα εμπορικά θέματα. Από εκεί έλκεται η προσωπική μου θέση σε αυτό το θέμα για τις λεπτομέρειες. Βλέπω στις τροπολογίες του το εισηγητή την 3, στην αιτιολογική σκέψη 3, ότι έχει διαγράψει το κείμενο της Κομισιόν. Η Κομισιόν θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανθρωπιστικός μέσα σε εισαγωγικό τρόπος για τη μείωση του πληθυσμού με φώνευση για τις φώκες. Η δική μου άποψη είναι ότι συμφωνώ με την Κομισιόν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ανθρώπινος μέσα σε εισαγωγικό τρόπος για να φωνεύονται οι φώκες και αυτό το είχαμε λάβει υπόψη όταν εγκρίθηκε αυτός ο κανονισμός το 2007. Η τότε η συνένεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος εξόντωσης ο οποίος να είναι ανθρωπιστικού χαρακτήρα και μας είχε, ε, το είχε διαφυσβητήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου τότε. Η ομάδα μου υποστηρίζει την εξαίρεση για τους Ινουίτ. Για μένα πρόκειται για να δοθούν οι δυνατότητες σε αυτήν την κοινότητα να επιβιώσει, όχι μόνο να έχει τροφή, αλλά να έχει τη δυνατότητα κάποιου εισοδήματο. Πιστεύω ότι αυτή η εξαίρεση θα πρέπει να είναι στο δυνατόν ευρεία για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η επιβίωση τη κοινότητα αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα για την εξαίρεση, σε ό,τι αφορά την διαχείριση των θαλασσίων πόρων, αυτό είναι διαφορετικό γιατί αυτό ήταν κομμάτι μια συμβαστική ε, ε λύση που οδήγησε στην απαγόρευση και η απαγόρευση θα είχε πάρει πολιτική υποστήριξη χωρίς αυτό το συμβιβασμό. Αν θυμηθούμε τι έγινε πριν από 7 ή 8 χρόνια. Αλλά είναι σαφής η απόφαση του ΠΟΕ λέει ότι αυτή η εξαίρεση θα πρέπει να αρθεί. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν να ρωτήσω τον εισηγητή είναι αν έχουμε περιθώριο ελιγμών εδώ μένοντα πάντα μέσα στου κανόνε του ΠΟΕ. Αλλιώ πρέπει να σεβαστούμε του κανόνε του ΠΟΕ, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε περιθώριο ελιγμών υπάρχει. Και η άλλη μου ερώτηση που είναι περισσότερο ερώτηση προς την Κομισιόν είναι πώς θα ασκήσει η Κομισιόν της εξουσίας της για εμπορικού χαρακτήρα θύρευση ώστε να μην υπάρχει ε, κατάχρηση των εξαιρέσεων γιατί υπάρχουν προβλήματα στην παρακολούθηση και την εποπτεία από ό,τι είδα σε τεχνικές συνεδριάσεις και γενικά εγώ υποστηρίζω τα σχόλια που έγιναν για τις πληροφοριακές εκστατείας με την προϋπόθεση ότι μπορεί να μείνει ως το δυνατόν πιο μικρός ο προϋπολογισμός μας. Θα πρέπει να ξέρουν όλοι ότι τα προϊόντα τα οποία έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αυτής της εξαίρεσης είναι νόμιμα. Αυτές λοιπόν θα είναι οι προτάσει που θα υποβάλουμε εμείς και εγώ προσβλέπω σε συνεργασία με τον εισηγητή και του άλλου κοιόδη εισηγητέ για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Ντόλτον. Από τη φιλελεύθερη ομάδα τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή έκθεσή του, το σχέδιο έκθεσής του. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τον εισηγητή για την συνεργασία του και το γεγονός ότι ήρθε, με, ήρθε σε επαφή με εκπροσώπους από το Κοινοβούλιο της Δανίας και της Γρυλανδίας. Ο εισηγητής ζητάει σχόλια για το σχέδιο έκθεσής του. Νομίζω ότι μπορέσατε να βρείτε μια καλή ισορροπία εστιάζοντας το πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη την απόφαση του ΠΟΕ και να συμμορφωθούμε με αυτή την απόφαση ενώ συγχρόνως σεβόμαστε τις εξαιρέσεις, ιδίως την εξαίρεση για τους Ινουίτ. Τούτου λεχθέντος όμως μας ε, ζητάτε την απόψή μας για την εξαίρεση MRM και δεν νομίζω ότι καλύπτεται απόλυτα αυτό το θέμα στο σχέδιό σα. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει πιο στεναρή διατύπωση για το θέμα αυτό. Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο η εξαίρεση MRM θα πρέπει να ε, απαλληθεί τελείως ή θα πρέπει να παραμείνει. Για μένα είναι ε, κάτι το οποίο είναι παράλογο. Μπορεί κανείς να θυρεύει φώκες στην Βαλτική, αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να μην χρησιμοποιηθεί η φώκια, αλλά να απορριφθεί και πάλι όταν έχουμε εγκρίνει μια πλήρη ε, απαγόρευση της απόρριψης θαλασσίων ειδών. Η εξαίρεση λοιπόν αυτή, η εξαίρεση για τη διαχείριση θαλασσίων πόρων, είναι τμήμα της ε, γνωμοδότησης και θα ήθελα και εμείς να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Όπως σας είπα, βρίσκω την, ε, ε, την εξαίρεση για τους Ινούιτ ότι είναι πολύ καλή και με τις απόψεις που ανέφερε ο εισηγητής για τον πολιτισμό, των Ινούιτ και την θήρευση των φωκοειδών. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα. Και θέλω να υποστηρίξω αυτό που έχετε στην έκθεσή σας σε σχέση με την εκστατεία συνειδητοποίησης του κοινού και την πληροφόρησή τους. Βέβαια αυτό δεν είναι για να κάνω κάποια διαφήμιση σε σχέση με τα προϊόντα από αλλά για να αποφύγουμε τις παρανοήσεις οι οποίες μπορεί να ισχύουν τις παρεξήγησεις που, νιώθουν, που τρέχουν πολλοί Ευρωπαίοι που θεωρούν ότι τα δέρματα από φώκες είναι απόλυτα απαγορευμένοι και με τον τρόπο αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτές τις παρανοήσεις. Και αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος της εκστατείας αυτής της πληροφόρησης. Είναι πολύ θετικό επίσης το ότι ο εισηγητής υπογραμμίζει το ότι η Κομισιόν υποχρεωμένη να δει τον αντίκτυπο αυτού του κανονισμού γιατί ελπίζω ότι όλοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλη είναι η επίδραση που μπορεί να έχει αυτή η απαγόρευση και οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινότητα των Ινουίτ, ιδίως στην Γρυλανδία. Είναι λοιπόν απόλυτα απαραίτητο να υπάρξει αυτή η ε, έκθεση αντικτύπου για τον κανονισμό. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το πολύ καλό έργο του και προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία μαζί του και με τους άλλους κοιόδης βέβαια. Σας ευχαριστώ και τώρα να δώσουμε το λόγο στους πράσινους, γιατί δεν νομίζω ότι είναι εδώ κανείς από τους ε, κοιόδης. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Βεβαίω και θέλω πάρα πολύ θετικό το θέμα της καλονταχύρισης των ζώων, το οποίο ελήφθη υπόψη ξεκάθαρα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει καλός τρόπος να σκοτώσει κανείς μια φόγια. Όμως, επισύρω την προσοχή σας και ζητά σας ευχαριστώ για το έργο σας, ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την ε, τροποποίηση του κανονισμού επειδή αυτό μας θέλει ο ΠΟΕ ούτως ώστε να ξεκινήσουμε την συζήτηση πάλι και έτσι να ξεκινήσει μια καινούργια στάθμιση διάφορων μεταβλητών της προβληματικής γιατί από πλευράς των πρασίνων ο ΠΟΕ Δύο θέματα μόνο θέτει για δύο παρεκκλήσεις. Στη μία ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις, ε, τους αδάσιους πόρους. Δεν χρειάζεται εδώ να γίνει κάποια εξαίρεση, οπότε λέμε ότι και η Επιτροπή σε αυτό και για τους Ινουίτ ομόφωνα θεωρούμε ότι αποκλείεται να τους θίξουμε τον τρόπο που έχουν για να υπάρξουν. Είναι αυτονόητο. Είναι θέμα ανθρωπισμού. Όμως, όπως λέει και ο ΠΕ, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως λέει και η έκθεση, θα πρέπει εμείς να βρούμε μια λύση που να εξισορροπεί την ε, ε, ύπαρξη του λόγου αυτού και το πώς θα ρυθμιστεί το εμπορικό κομμάτι. Οπότε και εμείς θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη στο πλάι του εισηγητή να δούμε πού θα καταλήξει ένα θεώρηση χρονισμού σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της ε, απαγόρευσης και μιας και μόνο εξαίρεσης υπέρ των Ινουίτ. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. EFDD. Μάρκο Τζούρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή. Εμείς φυσικά και συζητούμε με την πρόταση του ότι θα πρέπει να κατοχυρωθεί αυτή η απαγόρευση για τα προϊόντα φώκες. Και κύριε εισηγητά, αυτή η εμπορία είναι μια εμπορία βάρβαρη. Αυτό δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς. είναι βάρβαροι όσον αφορά το από πού παίρνουν το υλικό τη πρώτε ύλε, όσον αφορά τη βία που παιρνουν το υλικο τη πρωτη υλη οσον αυτή η πρακτική, ούτω ώστε να φωνεύσουν τι φωκέ. Είναι τρομερό να βλέπουμε εκεί πέρα τα, τα μωρά τη φώκια να, ε, να βρίσκονται σε πιθανά αγωνία που τα καρφώνουν, τα μαχαιρώνουν, τα, ξεκυλιάζουν ζωντανά. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία σε αυτόν τον κανονισμό. Γιατί σε κάποια κοινωνία πολιτισμένη δεν είναι δυνατόν αυτή η συμπεριφορά να είναι ανεκτή. Επίση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτά τα προϊόντα πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιούνται ε, μέσα από λαθρεμπορία. Και πρόκειται εδώ για περιπτώσεις απάτης, για περιπτώσεις οργανωμένου εγκλήματος. Οπότε γι' αυτό και θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν τόσο ώστε τέτοιες πρακτικές να σταματήσουν και να ε, τους προσάψουμε ένα αξιόπινο. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε εδώ, τελειώσαμε τώρα τους ε, σκιώδους γιατί είναι πάρα, πάρα πολύ ε, τυχερό το ότι έχουμε τώρα τον επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας για την περιοχή αυτή τον κύριο Ντόναν. Οπότε θα μα πει πώ έχουν τα πράγματα όταν μα εκπροσωπούσαν. Εκεί στο Δυτικό Σκανδιναβικό Συμβούλιο, που, τότε που υπήρχε η διακοινοβουλευτική συνάντηση τον Μάρτιο. Πολύ σημαντικό ότι χτε συζητήσαμε για τον ΕΟΧ. Όχι, τη Δευτέρα έγινε αυτό. Οπότε, να, πώς, πώς έχει σχέση με αυτά η Επιτροπή της οποίας προεδρεύεται. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πάρω το λόγο να θα μιλήσω εδώ στην Επιτροπή σας. Το θέμα θα απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλά μέλη και προκαλεί μεγάλη παρανόηση, όπως ε, ακούσαμε πριν από λίγο, για το πώς ε, γίνεται η θύρευση της φώκιας. Σας ευχαριστώ όμως για την ευκαιρία αυτή να σας παρακαλούσω τα αποτελέσματα της 27ης Μαρτίου της ε, κοινοβουλευτικής αυτής ε, συνέλευσης ε, που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες και περιλάμβανε ανταλλαγή πληροφοριών για τις τελευταίες εξελίξεις στα τρία μέλη του Σκανδιναβικού Συμβουλίου Ορλανδία, Ισλανδία και Ισδονίας. Το θέμα που συζητήθηκε ήταν η σύρευση της φώκιας και σχετική απόφαση του ΠΟΕ και σε σχέση με τις αλλαγές του κλίματος. Το θέμα της παραγωγής ε, προϊόντων φώκιας. Να σας πω ότι η Γρυλανδία υποσταρίζει και υποστηρίχθηκε από τις νήσες Φερόες για την κανονισμό του 2009 σε ό,τι αφορά την απαγόρευση τέτοιων προϊόντων στην εξαγωγή της τουλάχιστον και με τον εκκληστικό κανονισμό του 2010 οι δύο αυτοί κανονισμοί είχαν πραγματικά πολύ σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για του Ινουίτες στη Γλανδία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η αγορά για προϊόντα φώκιας πραγματικά έχει καταρρεύσει. Παρά όλα, παρά όλους τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις που έχουν εισαχθεί, η Γρυλανδία και οι νήσες Φερόε μας υποθύμησαν ότι τα προϊόντα αυτά αποτελούν σημαντικό τμήμα της ε, επιβιωσή τους και ότι το η θύρευση γενικότερα αποτελεί τη σημαντικό τμήμα της κουλτούρας τους. Δεν υπάρχουν, ξέρετε, στην Αρκτική ε, πολλά θελαστικά. Εδώ έχουμε βόλιο κρέα, έχουμε αυτονία, αλλά στον Αρκτικό κύκλο είναι περιορισμένα τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν στην ε, Ευρώπη επικρατεί μια αρνητική εντύπωση για τον αρχιπτικό κύκλο. Πρόκειται για ένα, μια κανονική μορφή θύρευση και οι μέθοδοι για την θανάτωση των ζώων είναι οι συνήθει. Ο εκπρόσωπος της Γρουλανδίας επίσης εξέφρασε την ιδιαίτερη ανησυχία για τις επιπτώσεις της απόφασης του ΠΟΕ που προτάθηκε από τον Καναδά και υποστηρίχθηκε από την Ορβηγία. Εμείς οι από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείναμε η Ιρλανδία να επιμείνει σε τρία σημεία στι συνομιλίε στα διεθνή φόρα, οι διάφορε μέθοδοι θύρευση φώκια, κατά δεύτερον το σεβασμό για την εξισορρόπηση των φυσικών πόρων και τον διαχωρισμό της στήρευσης φωκιάς στη Γρυλανδία σε σχέση με τον Καναδά. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός. Γιατί φαίνεται ότι μπλέκεται και η όλη συζήτηση για την επιλεκτική αλίευση. Το σημείο 2 και 3 στην διάταξη για τη συνεργασία και την ε, τον κανονισμό για το κλίμα. Χαίρομαι που εδώ ήταν συγκλίνους ε, οι απόψεις μας ε, μεταξύ Σκανδιναβικού κύκλου και Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δύο πιστεύουμε ότι η συνάντηση του Παρισιού το Σεπτέμβριο για το κλίμα θα πρέπει να προτιμαστεί σωστά και η Αρκτική είναι η περιοχή η οποία πλήττεται πιο έντονα από τι αλλαγέ στο κλίμα. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ όλοι. Πρόεδρο, και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Νίλσεν τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο συμβαίνει πολύ κοντά μας σε σχέση με τις φώκες και το θέμα της διατήρησης των θαλασσίων πόρων. Εγώ είμαι ιδιαίτερα επιθετικό για το γεγονό ότι η Κομισιόν έχει κοφεύσει στα συμφέροντα των σκανδιναβικών χώρων. χώρων. Καμιά προσπάθεια δεν έχει γίνει για να μπορέσει να συμβιβαστεί αυτό με τον, την απόφαση του ΠΟΕ. Φυσικά πρέπει να διατηρηθεί αυτή η συμφωνία, αλλά υπάρχουν ειδικέ καταστάσει για μα στη Βαλτική. Η αλίευση φωκών στην Βαλτική έχει σαν στόχο τη διατήρηση των θαλασσίων ειδών και την ε, διατήρηση των αλλιευτικών ε, πόρων. Περίπου 32.000 φώκες είναι εκεί και θυρεύονται στην Φιλανδία. Ίσως 500 στη Φιλανδία, 300 στη Σουηδία και άλλες 50 αλλού. Υπάρχει υπερπληθυσμός των φωκών, ο οποίος αυξάνεται και ασκεί πίεση στα αλλιευτικά ε, από θέματα στην Βαλτική υπάρχει έλλειψη ισορροπίας σε ό,τι αφορά την διαχείριση αυτών των φυσικών πόρων. Και όλα αυτά που γίνονται λοιπόν δεν το να μην υπάρχει θύρα των φωκών δεν συνάδει με την αλλιευτική μας πολιτική που πρέπει να βασίζεται σε αηφόρα αλλιεύματα. Το να ξεπεράσουμε αυτή την εξαίρεση καταρχήν εδώ πρόκειται για ένα θέμα θύρας που είναι μέσα στα εθνικά ε, κυριαρχικά θέματα, εθνική αρμοδιότητα. Είναι επίσης τελείως ανήθικο να κυνηγούμε τις φώκες οι οποίες μετά απορρίπτονται. Κανένας κυνηγό δεν θέλει να συμμετάσχει σε τέτοιες ενέργειες. Ελπίζω λοιπόν θα μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή λύση για το θέμα αυτό, γιατί αυτό το οποίο θέλουμε είναι να υπάρχει η διατήρηση εξαίρεση για τη διαχείριση φυσικών πόρων στην απόφαση εμείς όταν είχαμε κάνει αυτή την πρόταση βασιστήκαμε σε μία ε, νομική ανάλυση με συνεργασία των κυβερνήσεων της Σουηδίας και της Φιλανδίας και της Εστονίας. Ορισμένοι είπαν ότι αυτό ήταν απλώς ένας ελιγμός. Μάλλον ότι υπάρχει περιθώριο ελιγμών, αλλά η Κομισιόν δεν προσπάθησε να τον ε, εκμεταλλευτεί, να εκμεταλλευτεί αυτό το περιθώριο ελιγμών. Πρέπει να διατηρηθεί όμως η απόφαση του ΠΟΕ και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μην έρθουμε σε σύγκρουση με τον ΠΟΕ. Αλλά εγώ δεν συμφωνώ με την πρόταση της Κομισιόν ότι θα πρέπει να έρθει η εξαίρεση για την Βαλτική σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των θαλασσιών πόρων. Ξέρω ότι η Κομισιόν επίσης δεν προσπάθησε να δικαιολογήσει αυτή την εξαίρεση επί τη βάση των άρθρων του ΓΚΑΤ για την προστασία των φυσικών πόρων, αλλά προσπαθεί να αναφερθεί μονάχα στη δημόσια ηθική. Η Σκανδιναβική εξαίρεση λοιπόν θα πρέπει να διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η φώνευση ε, ε, φώνευση φωκών παρά μόνο για τη διατήρηση των αλληλευτικών ε, αποθεμάτων. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξουν ρήτρε εποπτείας όπου η Κομισιόν θα πρέπει να προβαίνει σε μια ανάλυση αντικτύπου τη θύρα για τις φώκες και τους αλληλευτικούς πόρους. Πρέπει να σεβαστούμε λοιπόν την απόφαση του ΠΟΕ, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια ρύθμιση των αποθεμάτων και όπου τα ζώα τα οποία φωνεύονται δεν θα απορρίπτονται, αλλά θα αντιμετωπίζονται σωστά. Χρειάζεται λοιπόν μια προσεκτική διαχείριση όλων αυτών των πόρων. Ευχαριστώ. έχω την Κομισιόν και ίσως θα είναι χρήσιμο να ακούσουμε την Κομισιόν. Οι DG Trade και DG Envin εμπλέκονται, ο Μάρτιν, Λούκας και ο Χάν Τιλστρο. Σας δίνω το λόγο. Thank you very much, uh, Madam Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε δύο λόγια για το πώς βλέπουμε την υλοποίηση των αποφάσεων του ΠΟΕ και μετά να προχωρήσουμε σε κάποια θέματα σχετικά με την εξαίρεση MRM και την εξαίρεση για τους Inuit. Όσον αφορά την προσάγγιση στην εφαρμογή της απόφασης, χειρουργική, περιορισμένη. Δηλαδή, να άρουμε όλες τις ε, ασάφειες και τις ασυνήπειες. Για τρεις λόγους. Πρώτον, θα πρέπει να τηρήσουμε την αυστηρή προθεσμία. Ζητούν μέχρι τον Οκτώβριο να έχουμε κάνει αυτό που αναλάβαμε. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θεωρηθεί ότι σέβεται τις υποχρεώσεις της. Επίσης, δεύτερον, αυτό είναι μια και έξω. Αλλά θα πρέπει κανείς με τη μία να πετύχει στην εφαρμογή όσον αφορά την απόφαση. Δεν μπορεί κανείς να ξαναπροσπαθήσει. Και τότε θα συρθεί ξανά ενώπιον του ΠΟΕ. Και γι' αυτό εξηγεί γιατί προετοιμαστήκαμε τόσο καιρό, θα πρέπει να κάνουμε διαβουλεύσεις για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια σωστή και ισορροπημένη πρόταση. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι όλα αυτά προέρχονται από δικαστική διαμάχη. Πρέπει να επερμηθούμε του κεκτημένου, κατόπιν να δούμε τις εξαιρέσεις και να δούμε αν θα πετύχουμε την απαγόρευση αλλά όχι για τις ε, εξαιρέσεις. Αυτά. Αλλιώς δεν θα ήμασταν συνεπείς με τα όσα είπαμε στην ε, Γενέβη. Δεν θα έχει νόημα επομένω η πολιτική μας. Τώρα, δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τέτοια περιορισμένη χειρουργική σύμφωνα για να υλοποιήσει τις αποφάσεις του ΠΟΕ. Πριν από μερικά χρόνια πριν, οι Κινέζοι είχαν προσβάλει τον κανονισμό για τον ντάμπινγκ. Και είχαν την ίδια προσέγγιση. Μόνο τροποποίησαμε μια διάταξη εκεί που πέτυχαν στην προσφυγή τους οι Κινέζοι. Τίποτα άλλο. και δεν έγινε και μελέτη επιπτώσεων γιατί αυτό είναι ε, ένδικη διαδικασία οπότε εμεί πρέπει να λύσουμε μόνο από τη βάση αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστούμε τον εισηγητή γιατί συμφώνησε με την προσέγγιση όπως λέει και το κείμενό του. Τον ευχαριστούμε. Πολύ σημαντικό για να συμμορφωθούμε με τον ΠΟΕ. Το για το MRM, με τις δύο εξαιρέσεις. Προτείνεται η κατάργηση της ε, εξαίρεσης MRM και η τροποποίηση της εξαίρεσης για τους Ινουίτ. Η διαφορά βγαίνει απευθείας από την απόφαση του ΠΟΕ. και είπε ο ΠΟΕ για την απαγόρευση σε σχέση με την καλοτοχή των ζώων δεν είναι δυνατόν να έχουμε εξαίρεση για κάποιο κυνήγι και να μην έχουμε εξαίρεση για ένα άλλο κυνήγι το εμπορικών σκοπών γιατί ακριβώς ε, απλώς δεν ε, δίνει μεγάλο κέρδος. Αυτό δεν είναι θεμητό λόγος για να υπάρχει διάκριση μεταξύ των δύο κυνηγιών. Η κυνηγούν διαφορετικά όπως ακούσαμε. Είναι θέμα ύπαρξης της κοινότητας των αυτοχθόνων οπότε αυτό θέμει επιχείρημα. Δεν είπαμε ότι το κυνήγι κατά τα λοιπά ε, είναι αχρίαστο, είναι σημαντικό και απλώς διαχείριση των πόρων. Αλλά σε περίπτωση απαγόρευσης να επιτρέψουμε κάποια προϊόντα να απολύονται από εκεί, αλλά όχι από άλλο κοινή γι' Αυτό είναι δεσμενή διάκριση. Εδώ στήθηκε ο ΠΟΕ. Οπότε και προσπαθήσαμε να τα επαναδιατυπώσουμε. Να σταματήσει η διάκριση και ταυτόχρονα να μην ε, υπονομεύσουμε την απαγορευστή, ένα δίλημα. λόγω του είδους εξαίρεση. Και τώρα η σκητάλη στον συνάδελφο για την άλλη εξαίρεση. Σας ευχαριστώ και εγώ από δικής μου πλευράς. Ε, να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε, που μας δώσατε την Επιτροπή, Τι που μας δώσατε το λόγο. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο σε σχέση με την έκθεση των εισηγητή. Να σας ευχαριστήσω που ακολουθείτε την λογική με αυτή που προσπαθούμε να προτάξουμε και στην πρόταση μας. Να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε δηλαδή την νομοθεσία με την απόφαση του ΠΟΕ. Η απόφαση του ΠΟΕ λοιπόν θα επικεντρωθώ σε αυτό το τμήμα της απόφασης. Μας έχει δώσει πολύ περιορισμένο περιθώρια για να διατηρηθεί αυτή η εξαίρεση IC. Το πολεμήσαμε και διατηρήσαμε αυτή την ευρότητα. Θέλουμε λοιπόν να την αξιοποιήσουμε. Γιατί, όπως είπαν και πολλοί άλλοι, θεωρούμε ότι αποτελεί ένομο συμφέρον της κοινότητας των Ινουίτ. Να κυνηγούν φώκες, και να γνωρίσουμε ότι αποτελεί αυτό αναπόσπαστο τμήμα της ταυτότητας και της κουλτούρας τους και σημαντικό για το βιός τους. Έχουμε βάλει λοιπόν στην νομοθεσία εκ νέου ένα μηχανισμό τον οποίο θεωρούμε αποδεκτό. Θεωρούμε ότι θα γίνει αποδεκτός από την απόφαση, βάσει του ΠΟΕ. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να είναι χρήσιμος και να εφαρμόζονται από όλη την κοινότητα των Ινουίτ στον Καναδά είτε στην Ιρλανδία. Καλασορίζουμε αυτά που είπε και ο εισηγητής σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση. Είχε την αίσθηση ότι εκ των υστέρων δεν θα έπρεπε να αποτελεί τμήμα της πρότασης. Υποστηρίζουμε τους λόγους τους οποίους ανέφερε το θέμα είναι ότι αν τώρα κάτσουμε να επανασχεδιάσουμε τον κανονισμό για τις φώκες προκειμένου να είναι συμβατός με την απόφαση του ΠΟΕ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσέξουμε προκειμένου να μην δημιουργηθεί κατά λάθο κάτι το οποίο θα προκαλέσει διακριτική μεταχείριση στη συνέχεια. Καλώς ορίζω λοιπόν αυτά που είπε ο σε σχέση με αυτό και έτσι λοιπόν κύριε Πρόεδρε, εδώ θα ήθελα να κλείσω. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή μας τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σύντομα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια. Φυσικά θα περιμένω για τις ε, ιδέες τους, για τις προτάσεις καλύτερης διατύπωσης ώστε να γίνει πιο σαφής η, θέση αυτή, η διατύπωση. Εγώ υποστηρίζω την ε, γενική άποψη ότι δεν χρειάζεται να ανοίξουμε και πάλι τη συζήτηση για ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί ήδη στο παρελθόν. Απλώς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας με την απόφαση του ΠΟΕ και να μην δημιουργήσουμε νέες διαμάχες νομικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να είμαι πάρα πολύ σαφές, πολλοί από τους ε, νομικούς συμβούλους με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή πιστεύουν ότι με τον τρόπο αυτό θα ανοίξει νέα διαμάχη σε νομικό επίπεδο. Εγώ υποστηρίζω την εξαίρεση για τους Ινουίτ όπως ελέγχθη και πιστεύω ότι είναι απόλυτα θεμητή η θύρευση από τους Ινουίτ και λαμβάνει υπόψη την ευζοία των ζώων. Θέλω ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι μας εξήγησαν την κατάσταση μετά την απαγόρευση και μετά το πέρασμα του βασικού κανονισμού. Είδαν ότι μειώθηκε το εμπόριο με τα προϊόντα φωκών γιατί πάρα πολλοί έμποροι στην Ευρώπη θεώρησαν ότι είναι παράνομο το εμπόριο αυτό και ήθελα να εξηγήσω ότι για τον πληθυσμό των Ινούιτ είναι νόμιμο κάτι τέτοιο και τα προϊόντα αυτά έχουν τη δυνατότητα να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε περιορισμένο χρόνο, μέχρι τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προετοιμάσει τις απαραίτητες νομικές πράξεις. Πρέπει να ψηφίσουμε λοιπόν τον Ιούλιο ή το αργότερα το Σεπτέμβριο. Είναι πραγματικά πολύ σφιχτό το χρονοδιάγραμμα, αλλά μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να τελειώσει εγκαίρως το χρόνο του να μπορέσει λοιπόν να συζητήσει μετά με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους και περιμένω ότι θα έρθουν οι προτάσεις σας για να με βοηθήσουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά, ευχαριστώ πολύ και τους και όλες η 20 Απριλίου είναι η καταληκτική προθεσμία. 7 Μαΐου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. 4 Ιουνίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας για να προλάβουμε την Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Θα ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και ευχαριστώ όλα τα μέλη. Θα ήθελα να σας πω ότι η επόμενη συνεδρία μας θα είναι στις 6 Μαΐου στις 9 το πρωί. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους κακόπαθημένους διερμηνείς.